Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί σήμερα έχουμε μία πολύ γεμάτη ημερήσια διάταξη, οπότε ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βαλτική και για τον ρόλο στην μελλοντική πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο εις τον εισηγητή να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του εγγράφου, τη γραμματεία, τους σκιώδης εισηγητές, Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την συνδρομή τους εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειών και εκ μέρους της επίσης όσοι συνέβαλαν από την Οικονομική και Πολιτική Επιτροπή. Υπάρχουν διάφορες ιδέες οι οποίες προέρχονται αυτή την τελευταία συζήτηση την οποία είχαμε κάνει. Αυτό που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές, οι μεταφορές και το περιβάλλον και ε, οι απόψεις είναι συγκλινόμενες με το έγγραφο όπου έχετε μπροστά σας. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ στα συμπεράσματα και μετά θα ασχοληθώ με την έκθεση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, διάφορες ε, προσπάθειες οι οποίες γίνονται και αν δείτε το πρόγραμμα ε, μεταξύ 2007 και 2013 αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μας απασχολεί και η πολιτική για τη Βαλτική καταρτίστηκε. Υπήρχαν και άλλες στρατηγικές για άλλες ε, ε, περιοχές ε, όπως είναι η Μεσόγειος και οι παραδουνάβιες χώρες. Τα θέματα αυτά συζητούνται στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Η στρατηγική για τη Βαλτική είναι πολύ σημαντική. Ε, ήθελε να ε, πρέπει να συζητήσουμε και για τις ανανεώσιμες πιές, ε, πηγές ενεργείας διότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία εις το να υπάρξουν συνεκτικές στρατηγικές ακόμη και στις μεταφορές γι' αυτό και εμπλέκεται η Επιτροπή Μεταφορών στην ε, περιοχή, σε διάφορες ε, περιφέρειες της περιοχής αυτής υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και το ίδιο ισχύει και για την οικονομική απόδοση. Ε, τα κενά αυτά λοιπόν πρέπει να ξεπεραστούν και η στρατηγική βασίζεται σε μία πολιτική συνοχής ε, σε σχέση με τις άλλες πολιτικές, παραδείγματος χάρη με την αλληλεία, με τις μεταφορές και όπως είπα και την κοινή ε, γεωργική πολιτική. Είναι επίσης πολύ σημαντικό και ε, συζητείται σε διάφορα ε, ε, σημεία διότι η στρατηγική για την Βαλτική αποτελεί μέρος μιας γενικότερης στρατηγικής ολοκληρώσεως της περιοχής και γι' αυτό βοηθάει και η μακροοικονομική στρατηγική για να μπορέσουν διάφορα περιβάλλοντα της περιοχής να ενταχθούν και η μακροπεριφέρεια πρέπει επίσης να ληφθεί, ε, περιφερειακή άποψη πρέπει να ληφθεί υπόψη, δηλαδή ε, το, ο τουρισμός, ε, η έρευνα, οι γνώσεις, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ή στην παιδεία και στην ακαδημαϊκή έρευνα διότι αυτά είναι στενά συνδεδεμένα με τη στρατηγική την οποία συζητάμε στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για ένα τεχνικό θέμα, πρόκειται για κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και ε, γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τα προβλήματα αυτά αυτά. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης της μακροπεριφερειακής προσέγγισης και ένα μέρος αυτής της χρηματοδοτήσεως προέρχεται από κάποια άλλα ταμεία, παραδείγματο χάρη το Ταμείο Συνοχής, όπου ορισμένες χώρες εμπλέκονται πολύ ενεργά. Είναι λοιπόν αναγκαίο να κάνουμε μία ανάλυση για το, τη μελλοντική μορφή που θα πάρει αυτή η ενίσχυση και θα δείτε στην παράγραφο 21 ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία αναφέρονται εις ε, ε, το σημείο αυτό και ε, θα το συζητήσουμε στο, τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Μπαστινάρου είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Ολένετσεκ για την εξαιρετική εργασία που έκανε. Η έκθεση είναι συνεπής, είναι ενδελεχής και ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη όλα τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας και άλλες μελλοντικές μικροπεριφερειακής ε, φύση. Ε, λόγω του γεγονότο ότι είμαστε η αρμόδια από τη ουσίες επιτροπή που ασχολείται με αυτή την έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά. Καταρχήν, όπως ήδη έχω πει και στο παρελθόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των ε, μη των κρατών που δεν ανήκουν στην Ένωση στι στρατηγικέ τη μικροπεριφερειακή ανάπτυξη. Δεν βλέπω δηλαδή πώ αυτέ οι στρατηγικέ θα μπορέσουν να εφαρμοστούν πλήρω και πώ θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του τη στιγμή που οι παίκτε, οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέλη τη Ένωση, δεν θα είναι ούτε και στο μέλλον μέλη τη Ένωση, αλλά έχουν ε, αντίκτυπο στι περιφέρειες για τι οποίε εμεί σχεδιάζουμε στρατηγικέ. Πώς λοιπόν μπορούν τέτοιου είδου στόχοι να επιτευχθούν χωρίς τη δική του συμμετοχή. Και μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, δεν σχετίζεται με κράτη της Ένωσης. Όπως ίσως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της ειδικής προεδρίας, η κυρία Μάλστρομ μας είπε ναι, το Nord Stream που υπάρχει στην έκθεση του κυρίου Λένιτζεκ είναι ακόμα ένα εμπορικό project, τίποτα παραπάνω. Όμως, εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργό της Ρωσίας, κύριος Πούτιν, ανακοίνωσε για το 2011 ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι απόλυτα λειτουργικό. Πολύ ωραία. Αλλά ο ρόλος της του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου πού βρίσκεται τώρα μετά την συνθήκη της Λισαβόνας μάλιστα όπου η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι εκτμήμα των κοινοτικών πολιτικών και εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω πως Αυτά τα προγράμματα έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν μιλάμε μόνο για την αυσιπλοεία και τις μεταφορές θαλάσσια στη Βαλτική θάλασσα, αλλά μιλάμε και για την ασφάλεια και άλλες τέτοιου είδους πτυχές. Και να αναφέρω και πάλι ότι πριν από δύο χρόνια, δύο επίτροποι, ένας που ήταν για το περιβάλλον, ο κύριος Δήμας, και ένας άλλος για την ενέργεια, που είναι τώρα υπεύθυνο για το περιβάλλον, ο κύριος Πίμπαλξ, μας υποσχέθηκαν ότι μετά από την έκθεση Λιμπίσκη για το Nord Stream θα υιοθετούνταν και μάλιστα υιοθετήθηκε τελικά με τεράστια πλειοψηφία μας υποσχέθηκαν λοιπόν πως η Κομισιόν θα ενημερώνει καταλήλως το Κοινοβούλιο για τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αξιολόγηση των επιπτώσεων σε αυτό. Είμαστε στις αρχές του 2010 και τίποτα δεν έχουμε δει σχετικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο και πάλι έχει μείνει στην πάντα, στην άκρη. Δεύτερη παρατήρηση. Τεράστια προγράμματα που σίγουρα θα έχουν ε, ε, επιπτώσεις και στη Βαλτική θάλασσα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα της μετώπισης καταστροφών. Τρεις καταστροφές που σχετίζονται με τεχνικά Συγγνώμη, είτε είναι για φυσι... πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για τρομοκρατικές επιθέσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια δραματική περίπτωση. Γιατί έχουμε ύδατα ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκά ύδατα, μη ευρωπαϊκά ύδατα και να πω και ότι έχουμε και αντινάτο ύδατα. Αλλά δεν έχουμε καμία στρατιωτική λύση σκεφτεί Πώς θα προχωρήσουμε σε τέτοιο δεχόμενο, θα πούμε στο ΝΑΤΟ, ε, περίμενε κύριε ΝΑΤΟ, έχουμε μια καταστροφή στη Βαλτική, δώστε μας την έγκριση για να μπούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ο ρωσικός τόλος θα πάει ή όχι. Κανείς δεν ξέρει σε τέτοια περίπτωση θα γίνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δραματική, όταν η αγωγή είναι τεράστια, δύο μέτρα φάρδο, ε, διάμετρο, ποιος θα πληρώσει την ύφη, σε περίπτωση ζημιάς. Γιατί αν δούμε και πάλι το εμπορικό, την εμπορική πτυχή και είμαι ευτυχής που είναι και τώρα α, επίτροπος η κυρία Μάλστρομ, αλλά ποιος θα πληρώσει την ύφη. Γιατί τίποτα μέσα στην εμπορική σύμβαση δεν αναφέρει τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό για να φτάσω στα συμπεράσματά μου να βάλουμε στις εταιρικές ε, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, Μολδαβία, Σερβία που σύντομα θα ε, μιλήσουμε και για τη στρατηγική του Δούναβη. Θα πρέπει να τοποθετούμε και όλα τα νομικά μέσα που σχετίζονται με την ε, βιοπικιλότητα και να, αποτελέσουν όλα αυτά τμήμα των κοινών μας νομικών διατάξεων για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προβλήματα. Και η, η, η Ρωσία υπέγραψε την ε, σύμβαση ΕΣΠΟ που είναι βασικό νομικό όργανο για το περιβάλλον αλλά ποτέ δεν επικύρωσε την σύμβαση αυτή την υπέγραψε μα δεν την επικύρωσε. Λοιπόν, είναι μια πρωτοπόρα έκθεση για οποιοδήποτε μικροπεριφερειακή συνεργασία και γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις για όλες αυτές τις ανησυχίες που έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Βίκτορ Μπαστινάρο. Τσέλερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ και είμαι ευγνώμων με τον κύριο Λινίτσα που κατήρτισε αυτό το έγγραφο εργασίας και του είμαι ευγνώμων και για την διαβούλευση την οποία είχαμε στην αρχή διότι είμαι σκιώδης εισηγητής για την πολιτική μου ομάδα. Ο προλαλής σας είπε ότι με την έκθεση αυτή που αναφέρεται στην μακροοικονομική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά και θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και αποφασιστικά πρέπει να είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προβεί στην μακροοικονομική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Γιατί το λέγω, διότι η μακροοικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να επιτύχει μόνο αν τα κράτη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή ε, εμπλακούν ενεργά. Είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση μιας τέτοια επιτυχημένη στρατηγικής και θα πρέπει οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα νησιά που βρίσκονται στην περιοχή να δραστηριοποιηθούν διότι περιμένουν πολλά από αυτή την ενέργεια αλλά προς το παρόν υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία διότι ε, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε και να θεωρήσουμε ότι τα κοινοβούλια τα οποία βρίσκονται στο χώρο της Βαλτικής πρέπει να κληθούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια. Διότι μόνο εάν μπορέσουμε ε, να συζητήσουμε όλους τους τομείς που αναφέρονται στην έκθεση ε, και συντονίσουμε τις πολιτικές αυτές θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και το βλέπω αυτό όσον αφορά ε, ε, το Κοινοβούλιο για τη Βαλτική ότι υπάρχουν ε, δύο εκθέσεις όπου υπάρχει αναφορά σε αυτή τη στρατηγική η οποία έχει συμφωνηθεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν πρέπει όμως αυτό να γίνει μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να είναι μέλημα όλων που εμπλέκονται στο χώρο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον χώρο και για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της Βαλτικής. Η εμπλοκή των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει ήδη θυγεί και νομίζω ότι τα προβλήματα δεν δημιουργούνται από τις διαμάχες για τις ακτές ε, της Βαλτικής αλλά αναφέρονται και στην ενδοχώρα χώρα και ε, τις, τις ε, γειτονικές χώρες οι οποίες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έχουμε επαφές με τα κοινοβούλια και τις συνελεύσεις αυτών των χωρών και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερο στη Ρωσία και θα πρέπει να συντονιστούμε. Θέλω όμως τώρα να έρθω σε ένα θέμα το οποίο ανέφερε πολύ ρητός ο προλαλής σας. Δηλαδή σχεδόν ε, σαν αντίδραση βλέπω ότι όποτε μιλάμε για στρατηγική της Βαλτικής ε, προκύπτει και τίθεται στην ημερήσια διάταξη το πρόβλημα Nord Stream. Το Nord Stream είναι μια πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Διότι την προηγούμενη θητεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κληθεί να καταρτήσει μια έκθεση το οποίο δεν έχει πράξει ακόμη και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν το έχει πράξει είναι δικαίωμά μας. Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για ε, περιβάλλον και προβλήματα επικοινωνίας και μεταφορών, το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί ε, να λυθεί παρά μόνο ε, αν ε, τα κράτη τα, της Βαλτικής μέσω των οποίων θα περάσει αυτός ο αγωγός συνενέσουν είναι δικαίωμα κυρίαρχο δικό τους και γι' αυτό θα πρέπει να καταρτήσουμε μία στρατηγική πολύ πιο εκτενή από ένα μεμονωμένο πρόγραμμα. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται πρέπει να λάβουν απάντηση, είναι σαφές, αλλά η στρατηγική της Βαλτικής είναι πολύ ε, πιο ευρεία από ότι μόνο την κατασκευή ενός αγωγού χρειάζονται και άλλα προγράμματα υποδομής ε, τα οποία χρειάζεται η περιοχή. Είναι θέματα που πρέπει να θυγούν και εκεί ε, το Nord Stream θα αποτελέσει μόνο ένα από τα θέματα και αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε είναι την καλύτερη διασύνδεση του βορειοανατολικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την υπόλοιπη κατά τρόπον ώστε ε, για τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές να υπάρχει καλύτερη μελλοντική προοπτική και ε, ιδίω ε, εφόσον ε, η Βαλτική έχει γίνει εσωτερική κοινοτική θάλασσα να μπορέσουμε να μειώσουμε τις πιέσεις που τις επιβάλλουμε. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε από αυτή τη σκοπιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε με τους κοιόδες συζητητές. Ρίκα Μάνερ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Όλα αυτά, ε, ε, αυτά είπαν, ε, υπόθηκαν ήδη από άλλους ομιλητές. Αυτή την έκθεση διαπιστώνουμε πως έχετε εμβαθύνει πολύ στο θέμα κάποιες παρατηρήσεις. Η στρατηγική αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική είναι, θα αποτελέσει μάλλον παράδειγμα και για άλλα τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και για το μέλλον είναι επίσης πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να μπορούμε να τα λειτουργήσουμε όλα αυτά από τη διοικητική άποψη και να έχουμε φυσικά και τα απαραίτητα κονδύλια που θα συνοδεύσουν αυτήν την στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρόγραμμα αυτό, αναφέρονται διάφορες προκλήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διοικητικά θέματα και τη διαχείριση ε, ίσως θα πρέπει να επιμείνουμε κάπως περισσότερο για την εφαρμογή αυτών των διαφόρων στοιχείων στο πλαίσιο αυτής της ε, μικροπεριφερειακής στρατηγικής. Δεν θέλουμε νέες δομές ή νέους οργανισμούς, γιατί έχουμε ήδη οργανισμούς υπάρχοντες. Άρα πρέπει να αναλάβουμε τη διαχείριση όλων αυτών μέσω της ε, αξιολόγησης, αξιοποίησης των υπαρχόντων ε, φορέων. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερο διοικητικά διοικητικούς φορείς. Αυτό θα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Οι δομές θα μας χρησιμεύσουν για να διοχετεύσουμε, να δρομολογήσουμε μάλλον τη χρηματοδότηση σε αυτό το τομέα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην συνεργασία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να εμπλέκει τα διάφορα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, ε, εθνικό και διεθνές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό αν θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πιστεύω επίσης πως κάτι ακόμα είναι ε, πολύ θεμελιώδου σημασίας, όπως είπε ε, και η συγγήτρια, ο εισηγητής, συγγνώμη, στην ε, εισήγησή του, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι έχει ήδη γίνει στο τομέα επιτόπου. Κάτι ακόμα σημαντικό, η βιοενέργεια, η παιδεία, η πολιτική γυπνίασης, όλα αυτά είναι στόχοι εξαιρετικά σημαντικοί για την, περιφε... για την ε, Βαλτική. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν όλα αυτά επί τόπου. Άλλο ερώτημα είναι πώς θα μεταφράσουμε στην πράξη όλους αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να βρίσκεται σε αυτό το έγγραφο, συχνά αναφερόμαστε στη στρατηγική 2020. Πρόκειται για στόχους τους οποίους βρίσκουμε στο εγγραφό αυτό και που συνδέονται με τη στρατηγική 2020. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος δεσμού σύνδεσης με αυτή τη στρατηγική 2020, δηλαδή ανάμεσα στους διάφορους στόχους και τη στρατηγική 2020. Στη συνέχεια, όπως είπε και κάποιος προηγούμενος ομιλητής, το πρόβλημα δεν τίθεται μόνο για την Βαλτική και τις όχθες της. Το πρόβλημα μπορεί να αφορά και το εσωτερικό των χωρών αυτών. Μιλάμε επίσης για την πολιτική της αιρτικής. Α μην ξεχνάμε πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, αρκτικές περιοχές. Ας τις λάβουμε υπόψη. Ας λάβουμε υπόψη την ε, βόρεια διάσταση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό αυτής της περιοχής. Θα ήταν καλό λοιπόν να αναλαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βόρειες αυτές τι περιοχές γιατί όπως σα το είπα εξαρτάται από αυτό το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Nord Stream τώρα. Το Nord Stream είναι μια πραγματικότητα για την Ευρώπη και για τη Βαλτική. Μιλήσαμε για την ε, μελέτη ε, αξιολόγηση των περιβάλλων. Αυτή έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο. Οι συμβάσεις ε, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ίσως λοιπόν σε αυτό το έγγραφο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη το γεγονός αυτό και να μιλήσουμε για θέματα ασφάλειας, πλοήγησης, τα κτλ. Ε, σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι με, ε, μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ο κ. Φρανσουά Αλφονσί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που έδωσε στην έκθεσή του μία διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα εφόσον τονίζει πέραν της Βαλτικής μία στρατηγική για την ε, περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη. Θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ε, θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις μεταφορές διότι παραδείγματος χάρη οι ε, θαλάσσιες ε, μεταφορές είναι πιο σημαντικές ε, και μόνο με τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της ευρύτερης περιφέρειας. Χρειάζεται δε να ε, αναφερθούμε ε, σε αυτήν την ιστορική λεκάνη της Ευρώπης ε, ε, όταν μιλάμε για το πρόγραμμα που εξετάζεται και τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί. Ε, υπάρχει ένα θέμα που μας απασχολεί για το μέλλον. Η επικουρικότητα όπως καταρτίζεται από την συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ σημαντική για να τονίσουμε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται για να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση και για τους χρήστες σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα καλύτερα επιτυχάνονται οι στόχοι σε επίπεδο ενώσεως από σε επίπεδο κρατών και αυτό που εμπλέκεται δεν είναι άμεσα τα κράτη Πρέπει λοιπόν να τονιστεί αυτή η ανάγκη αντιμετωπίσεως της επικουρικότητας και το λέγω αυτό διότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάπως το σημείο 19. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάπως επιφυλακτική και γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει μια στρατηγική η οποία να πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω. Εάν θέλουμε δηλαδή να υπάρξει μια στρατηγική ιστορική στις λεκάνες αυτές θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να έχουμε προβλέψει και τα εμπλεκόμενα κράτη να έχουν αρχίσει να σκέφτονται το θέμα αυτό και να προετοιμάζονται για να διατυπώσουν προτάσεις οι οποίες θα βασίζονται στη βάση και δεν θα προέρχονται από την κορυφή. Από τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσει τα μέσα που χρειάζονται για να βρίσκεται το θέμα αυτό στο επίκεντρο της δράσεώς της. Ευχαριστώ. Υπάρχει εδώ ο επόμενος ομιλητής, διότι διαφορετικά θα πάμε στον κύριο Όλμπριχτ. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Νομίζω πως ήταν η σειρά του εισηγητή για το ECR. Να κάνω κάποιες σύντομε παρατηρήσει. Πιστεύω πως αυτή η έκθεση, αφού μάλλον συγχαρώ τον κύριο Όλιντζεκ, δεν είναι κάτι το τυπικό. Ε, τυπικά τα συγχαρητήριά μου. Είστε νεοαφιχθεί και η ποιότητα της έκθεσής σας είναι εξαιρετική. Ε, η έκθεση αυτή είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί αφορά τη στρατηγική της Βαλτικής, αλλά πρόκειται για την μα, μικροπεριφερειακή στρατηγική μας για το μέλλον. Δηλαδή τα όσα πούμε τώρα θα έχουν συνέπειες για το μέλλον. Να σας θυμίσω πως μέχρι τώρα η περιφερειακή πολιτική η πολιτική συνοχής βασιζόταν σε υποεθνικό περιφερειακό επίπεδο ΝΑΤΣ 2. ΝΑΤΣ 2. Για το μέλλον ε, το θέμα είναι η πολιτική συνοχή. Θέλουμε να αλλάξει και να προχωρήσουμε πέρα από το ΝΑΤΣ 2 στο ΝΑΤΣ 1 ή θέλετε να μείνουμε στο επίπεδο ΝΑΤΣ 2 και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος περιφερειακής πολιτικής που θα αποκαλείται μικροπεριφερειακή πολιτική. Είναι πολύ στρατηγικό θέμα αυτό. Εάν θέλουμε να μείνουμε στο ΝΑΤΣ 2, τα χρήματα τα χρήματα θα πηγαίνουν στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους μετά θα συνεργάζονται. Αν θέλουμε να έχουμε μια νέα μακροοικονομική, μικροπεριφερειακή στρατηγική σημαίνει πως η στρατηγική ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ε, απέναντι στην μικροπεριφέρεια, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η στρατηγική συνεργασία, είναι η στρατηγική της Ένωσης που μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών ΜΚΟ. Εάν λοιπόν θέλουμε να συμπεριληφθεί η πολιτική σε έρευνα, αλληλεία και όλα τα θέματα αυτά, είναι το θέμα που μετά τίθεται ποιος θα τα συντονίσει όλα αυτά και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξεκινάμε με το Δούναβι. Κανείς εδώ δεν με το λέει, αλλά όλοι γνωρίζουν πως διάφορα κομμάτια της Ευρώπης ετοιμάζουν τέτοιου είδους περιφέρειες. Όλοι ετοιμάζουν τα, να, τα Πυρηναία, η Μεσόγειο, η, τα Καρπάθια. Θέλουμε δηλαδή να φτιάξουμε αυτή τη νέα μικροπεριφερειακή πολιτική ή θέλουμε να έχουμε προ... θέλουμε, ε, θεωρούμε μάλλον πως είναι προβληματικές αυτές οι περιοχές. Μήπως θα πρέπει να έχουμε μια νέα περιφερειακή σκέψη, να ορίσουμε την μικροπεριφέρεια, διότι αυτό είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, όπως αυτό που αφορά τη Βαλτική θάλασσα π.χ. Αλλά βέβαια σημαίνει ότι θα υπάρξει και επικάλυψη των μικροπεριοχών αυτών, γιατί θα γίνει ο χωρισμός επί τη βάση λειτουργικών διαχωρισμών και όχι γεωγραφικών παραδοσιακών γεωγραφικών διαχωρισμών όπως το μπασάν που λέμε στα γαλλικά η λεκάνη. Το να σκεφτούν από κοινού οι διάφοροι φορεί για τις κοινέ προτεραιότητε και ένα κοινό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό και έχει προστεθεμένη αξία. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε ως μια νέα πολιτική, μικροπεριφερειακή και βεβαίως αν θεωρούμε πως είναι μόνο πολιτική συνοχής, αυτό δεν έχει κανένα, καμία σχέση μετά με τον Nord Stream, γιατί η πολιτική συνοχής δεν έχει σχέση με τον Nord Stream. Αλλά αν πούμε ότι πρόκειται και αφορά όλες τις πολιτικές, φυσικά τότε εκεί μπαίνει και το Nord Stream, γιατί είναι πολιτικό θέμα, ε, περιβαλλοντικό, οικονομικό κτλ είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ακριβώ τι είδου πραγματικότητα είναι. Δεν θέλω να μπω να γράψουμε μέσα στην έκθεση ναι, ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα, γιατί θα αρχίσουμε να μιλάμε για οριστείες, για την εικονική, την πραγματική πραγματικότητα, την εικονική πραγματικότητα και το ούτω καθεξής. Αλλά κατά την άποψή μου στην έκθεση, η έκθεση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ σοβαρά, να ληφθεί υπόψη ως το πρώτο βήμα. Τι θέλουμε εμείς ως Επιτροπή. Θέλουμε περιφερειακή πολιτική, θέλουμε μια νέα περιφερειακή πολιτική, θέλουμε μικροπεριφερειακή πολιτική εντός του στόχου 3. Δηλαδή εδαφική συνεργασία, αυτή είναι η κύρια διαφορά. Δυστυχώς αυτή η έκθεση δεν κλείνει τη συζήτηση, την ξεκινά. Είναι το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Λέω ο και εγώ θέλω να έρθω για να συμφωνήσω με όσους πιστεύουν ότι εδώ δεν έχουμε μία περιοδική διαδικασία το να ακούμε και να ευχαριστούμε τους ε, εισηγητές γιατί με μεγάλη μου χαρά άκουσα ε, αυτά τα τόσο αξιόλογα που είχε να μας πει. Συμφωνώ 100% με αυτά που είπε ο συνάδελφος Άλμπριχτ. Τώρα έχει γίνει κάτι σαν παράδοση. όταν συζητάμε κάτι, κάτι σοβαρό, μιλάει πρώτα ο κ. και μετά εγώ όμως συμφωνώ 100% με αυτά τα οποία είπε και κατά τη γνώμη μου. Εδώ δεν έχουμε μία έκθεση, έχουμε δύο. Γιατί ξεκινάμε με ένα κομμάτι πάρα πολύ αξιολόγο το οποίο ασχολείται με την περιοχή της Βαλτικής και την υλοποίηση της ε, στρατηγικής, την αξιολόγηση της στρατηγικής και κατόπιν έχουμε και άλλη μια έκθεση η οποία αφορά τα θέματα που μας ανέφερε ο κύριος Αλμπριχτή δηλαδή. Τι θα γίνει με τις διάφορες εκεί περιφέρειες, τι θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρόκειται εδώ για μια πάρα πολύ αξιόλογη έκθεση που έχει το άριστο τμήμα και το πολύ καλό Οπότε συγχαρητήρια κύριε Άλμπρεχ και παρακαλώ έχω να πω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το δεύτερο τμήμα της έκθεσης. Μπορούμε να αρχίσουμε την ε, συζήτηση αλλά θα πρέπει αν μη τι άλλο να θέσουμε κάποια ερωτήματα σαν αρχή της συζήτησης. Διότι ξέρετε για πολύ καιρό είχαμε με αυτή την μονομαχία, την αναμέτρηση για το αποτέλεσμα. Και η μονομάχοι καθόντουσαν εκεί, κοιτούσαν στον τον άλλον, δεν σήκωναν το ξύφο του. Και έτσι το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Γίνεται αυτό πολλέ φορέ στην ξυφομαχία, ξέρετε. Αυτό σημαίνει και τώρα. Αναμονή για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών προοπτικών σε σχέση με την περίοδο 2013 για τα δημόσια οικονομικά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μικροπεριφέρειες και σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική. Οπότε, όλα εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Έτσι είναι ο κόσμος. Είναι αλληλένδετες αυτές όλες οι πράξεις αυτά τα φαινόμενα. Οπότε θα πρέπει να παραδειχτούμε ότι υπάρχει αυτή η αλληλουχία και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλα μαζί να τα σκεφτούμε. Αλλά τελικά κάπου να καταλήξουμε. Και με την έκθεση αυτή να μπορέσουμε τουλάχιστον να θέσουμε κάποια βασικά στρατηγικά ερωτήματα. Γιατί είμαστε Περιφερειακή Επιτροπή του Κοινοβουλίου και εμείς αλλά και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των μικροπεριφερειών. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να θέσουμε. Και το 66% αυτών τα έχει θέσει και ο Σάλμπουρτ και είναι επομένω σε αυτή η έκθεση δύο πάρα πολύ αξιόλογε θέσει. Ακριβώ, όπω είπε ο κ. Σόλιτσεκ, συνάδελφοι και από την Οικονομική Επιτροπή όπως και εμείς επεξεργαζόμαστε την έκθεση αυτή για να τα αναλύσουν τα θέματα αυτά με τους ε, εισηγητές μας. Τώρα έχουμε τρεις συναδελφούς που έχουν λάβει το λόγο και παρακαλώ περιοριστείτε στα τρία λεπτά ο καθένας γιατί στις 10 θα πρέπει να ψηφίσουμε. Όμως μετά από τους αγορητές θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ξεκινάμε. Το κ. Σμίθ από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ολέντζεκ διότι έχουμε τώρα την ευκαιρία ε, εδώ έχουμε μακροσκελής εκθέσεις όσον αφορά την μακροπεριφερειακή συνεργασία στην ε, Επιτροπή μας τα συζητάμε αυτά οπότε γι' αυτό και ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σημερινή έκθεση Έχουμε μια γενική ε, διατύπωση κριτικής, ε, είναι κάποια σχόλια θετικά για την, αυτή την μακροπεριφερειακή αντιμετώπιση, αλλά όπως σήμερα το πρωί ακούστηκε η στρατηγική για την Βαλτική επιδέχεται πάρα πολλές βελτιώσεις και έχουμε ένα σωρό θέματα τα οποία κρεμούν, είναι ανεπίλητα. Οι δε πολιτικές δυσκολίες είναι πιο μεγάλες από τις ε, οικονομικές. Και αναρωτιέμαι, γιατί αυτά δεν τα έκανε πιο πριν η Ευρώπη. Ίσως γιατί έχουμε τώρα περισσότερη ακαιρεότητα της Ευρώπης, περισσότερη ολοκλήρωση, μια που έχει γίνει η διεύρυνση. Οπότε να, γιατί αναδείχθηκε αυτή η μακροπεριφερειακή διάσταση όμως. Ε, δεν έχουμε πάντοτε ταύτιση των ε, πολιτικών εθνικών συνόρων με, τη, με τα περιφερειακά και επομένως κάποιες τέτοιε δύσκολε πολιτικέ και προβληματικέ δεν μπορούμε να τι εντοπίσουμε έτσι γιατί ακριβώ, ε, αυτά τα οποία ε, ισχύουν τώρα δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται στην πρόκληση. Η δε μακροπεριφερειακή προσέγγιση αυτή είναι η ιδεώδη λύση για να πετύχουμε το στόχο μα. Μην ξεχνάμε όμω ότι με τι στρατηγικές αυτές μακροπεριφερειακές αυτή τη στιγμή ξεκινάμε ένα πάρα πολύ μεγάλο τεστ και ένα πείραμα τόσο ώστε να μπορέσουμε αυτέ τι ε, ιδέε να τι μετασχηματίσουμε σε κάποιε πράξεις για το περιβάλλον, για ε, καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Και τώρα με ποιο σχήμα θα γίνει αυτό, με τι διακυβέρνηση. Ε, αυτά θα καθορίσουν το κατά πόσον θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να φέρουμε αυτές τις αλλαγές και να μπορέσουμε να δώσουμε προτεραιότητες εκεί που πρέπει και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση ξεκίνησε και γεννήθηκε σαν ιδέα εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο τώρα σπρώχνει προς την ε, εφαρμογή. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά και εγώ επομένως από πλευράς μου στην ΟΚΕ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω. Εμείς ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος και τώρα δώσουμε το λόγο στην ε, Παγωλίνα Χάιάνεν από την Επιτροπή των Περιφερών που είναι η εισηγήτρια για την αντίστοιχη έκθεση στην ε, Επιτροπή των Περιφερειών. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία, κυρίε και κύριοι. Να σας πω δύο λόγια για την στρατηγική αυτή από πλευρά της Επιτροπής των Περιφερειών. Για να συνεχίσω στη συμμετρική μου γλώσσα τα φινλανδικά. Για τη Βαλτική, επομένω, έχουμε αναλάβει αυτή την προσπάθεια, γιατί και ξεκίνησε αυτό με μια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου το 2006. Ξέρετε, πάρα πολλοί έχουν εμπλακεί, ούτω ώστε να μπει σε καλό δρόμο η τη Οπότε ε, θέλουμε να υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο να το ακολουθήσουν και άλλε μακροπεριφέρειες στο μέλλον. Οπότε γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι όλοι οι κλάδοι, όλοι οι όλα τα επίπεδα συντονισμένα έχουν εμπλακεί. Και ξέρετε, με την επεξεργασία αυτής της στρατηγικής η Επιτροπή επέμεινε στο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω και να πάμε προς τα πάνω, από χαμηλά προς τα ψηλά. Και εδώ έχουμε δύο στοιχεία που πριν ανέβουν και τα τονίζω αυτά στην δική μου έκθεση, στο δικό μου κείμενο. Πρώτα-πρώτα έχουμε την εξωτερική διάσταση της στρατηγικής αυτής και κατόπιν έχουμε το ρόλο της ε, τοπικής και περιφερειακής ε, διοίκησης. Οπότε για αυτή τη στρατηγική θα πρέπει κανείς να σταθεί στα ζητήματα που αφορούν πρώτα απ' όλα την εξωτερική διάσταση Ισλανδία, Νορβηγία και Ρωσία. Θα πρέπει και αυτές οι χώρες να εμπλακούν σε αυτή την συνεργασία για τη Βαλτική. Επομένως, θα πρέπει όλες αυτές οι περιφέρειες να συνεργαστούν. Αλλά και η Ουκρανία. Όλα αυτά επομένως θα πρέπει να θυγούν από την στρατηγική αυτή. Θα πρέπει να καλυφθούν και θα πρέπει επομένως σε κάθε επίπεδο να προχωρήσουμε, να επεξεργαστούμε τους στόχους που έχουμε θέσει και ο κάθε στόχος να συνδεθεί με κάποιο πρόγραμμα ε, συνεργασίας. Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την χρηματοδότηση που θα πικοδοτήσει αυτή την στρατηγική. γιατί αυτά τα προγράμματα ε, εμπλέκουν και την Ρωσία. Οπότε και εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι τώρα μιλούμε για μακροπεριφέρειες. Και η συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια που μας απασχολεί εν προκειμένου θα πρέπει να καλύψει όλες τις αρχές σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι θα πρέπει να γίνει αυτή η στρατηγική και να μην απομακρύνουμε, τους φέρουμε πιο κοντά τους Ευρωπαίους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει επομένω η, η εκεί αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή κάτι να κάνει ούτω ώστε να ελκύσουμε την ε, κοινή γνώμη για την ε, υπόθεση αυτή της στρατηγική της Βαλτικής. Τώρα, όσον αφορά την υλοποίηση της ε, στρατηγική. Όλα εξαρτώνται κατά πολύ από το πώς θα εμπλακούν και τρίτες χώρες στην υπόθεση αυτή. Και έτσι μόνο θα αστευτεί με επιτυχία το εγχείρημά μας. Νομίζω ότι πρόκειται εδώ για ένα όραμα πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο θα μπορούσε ε, μετά την πιλωτική αυτή φάση να ισχύσει και για άλλες μακροπεριφέρειες. Αυτά θα να σας τονίσω. Ευχαριστώ ε, και την εισηγητριά σας ή τον εισηγητή σας για την τόσο καλή ε, συνεργασία. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής από την Επιτροπή των Περιφερειών είναι ο κ. Αλτέγκρε που είναι εισηγητής για την ε, σχετική έκθεση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε σε αυτήν την συνεδρίαση. Λέγομαι Ναλγκέν, και είμαι μέλος της Επιτροπής Περιφερειών, αλλά επίσης και πρόεδρος της, ε, του Group Interbaltikis. Μιλάμε για τις μικροπεριφέρειες και τη Βαλτική θάλασσα ως μικροπεριφέρεια επίσης. Πιστεύω πως οι μικροπεριφέρειες στην Ευρώπη είναι ένα πολύ καλό συμπλήρωμα στην πολιτική συνοχή. Δεν πιστεύω πως μπορεί να υπάρχουν μικροπεριφέρειες ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά Υπάρχουν ε, λειτουργικές περιφέρειες όπου μπορείς να το κάνεις αυτό και αυτό το τμήμα της Ευρώπης είναι πολύ καλό να έχει μια τέτοια συμπληρωματική πολιτική συνοχή. Είναι σημαντικό η ε, διασύνδεση ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά επίπεδα που θα πρέπει να συνδέονται καλά εάν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει αυτή η πολιτική. Ο τρόπος για την ενσωμάτωση αυτών των πολιτικών είναι πολύ θετικός, έτσι όπως περιγράφεται σε αυτή την έκθεση. Θεωρούμε πως ε, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή για κάθε ένα από αυτά τα θέματα προτεραιότητας και εκεί καλούνται οι περιφέρειες να συμμετάσχουν, να εμπλακούν ε, ενεργά. Όσο περισσότερο ολοκληρωμένες είναι οι προσεγγίσεις, τόσο πιο αποτελεσματικές είναι. Ε, αυτή η στρατηγική βασίζεται στο περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και πιστεύω πως θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η βιώσιμοι ε, στόχοι δεν ε, μπορούν να επιτευχθούν ε, από μόνοι τους, εξαρτώνται από ολόκληρη την περιφέρεια και όλους όλη τη συνεργασία. Ε, τμήματα της κάθε περιοχής μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κάθε περιοχής αναλόγως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν συζητάμε τα θέματα ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, μπορεί να υπάρξει αντίφαση ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες και αυτό δεν βοηθάει για την ανάπτυξη στο μέλλον. Να πω και δύο λόγια σε σχέση με την ε, συνοχή, τη Ρωσία, την Νορβηγία και την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Είναι πολύ καλό νομίζω θετικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δική της ε, στρατηγική ε, μικροπεριφερειακά και θα είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με τη Ρωσία από την άποψη, την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε προσπαθήσει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία και τις διάφορες χώρες στην Βαλτική και θα... Ε, ε, κάποιες φορές έχουμε πετύχει, πάντως γενικά όχι. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει για την βόρεια διάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο λεπτά ο David Sweet. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διατηρεί ψηλά το επίπεδο του ενδιαφέροντος αλλά και της, του προβληματισμού και της πολιτικής όθησης για ολόκληρη αυτή την προσέγγιση. Γνωρίζουμε πως από εδώ ξεκίνησε η ιδέα και, πως, και πιστεύουμε πως αυτή η έκθεση είναι μια πολύ αξιόλογη συνέχεια. Ε, μακάρι να είχα χρόνο να αναφερθώ μεμονωμένα σε όλες τις ιδέες αυτές που ακούστηκαν σήμερα, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα πω μόνο τα εξή. Το πρώτο σημαντικότερο είναι ότι κατά πόσο αυτή η στρατηγική είναι ένα πρόγραμμα η ίδια, είναι είδος πειράματο, πιλωτικού προγράμματος. Είναι και τα δύο και θα πετύχει μόνο εάν ...κάνει τη ζωή καλύτερη στις περιοχές αυτές της Βαλτικής θάλασσας. Δεν είναι μόνο μια ακαδημαϊκή ε, προσπάθεια, ε, αλλά προσπαθεί να κάνει και τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές αυτές καλύτερη. Ε, και πολύ όπως σας το τονίσατε, αν μπορεί αυτή η υπόθεση να λειτουργήσει πιο καλά. Το κάναμε στην προηγούμενη επιτροπή, το γνωρίζει η Πρόεδρος η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει πολύ προσεκτικά πού μπορεί να πάει, ιδιαίτερα ε, ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε, γιατί πρέπει να έχουμε αποτελέσματα και δεύτερον ποιους πόρους μπορούμε να εφαρμόσουμε και ποιο είδος ε, ε, μηχανισμού χρηματοδότησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αναφερόμαστε στους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της Κομισιόν Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο περισσότερο input από την Κομισιόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε, ό,τι, ό,τι μας δίνουν θα το πάρουμε, διότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε τα αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε από τη Βαλτική και από το Δούναβη και κατά πόσο αυτό δικαιολογεί το να πάρουμε κόσμο από άλλους τομείς και να τους βάλουμε να εργάζονται για αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε με την ε, Κομισιόν. Επίσης το θέμα των εξωτερικών σχέσεων είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να σας πω ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά, ειδικά με τη Ρωσία, Έχουμε επαφές με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και το Υπουργείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. πολύ θετικές οι επαφές, πολύ πιο θετικές από ό,τι ελπίζαμε και υπάρχει κάθε προοπτική τουλάχιστον να υπάρχει μια κάποια ελευθερία για τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές τους ε, τοπικούς φορείς εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συμμετέχουν πλήρως προς το δικό του συμφέρον φυσικά στις διάφορες δράσεις που γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να προσβλέπουμε σε πιο στενή συνεργασία και κατανοώ τα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει, μας βρίσκουν σύμφωνους. Ε, καλωσορίζουμε την προσέγγιση, ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Επιτροπής σας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και ε, θα προσέξουμε κάθε προσπάθεια προετοιμασίας. Σας ευχαριστώ. Θα να πω πως όχι μόνο οι συγητής, αλλά και όλοι οι σκιώδεις που συμμετείχαν σε αυτήν την ε, πολύ ουσιαστική συζήτηση, να τους ευχαριστήσω. Έχουμε 24 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα προθεσμία ε, για υποβολή ε, τροπολογιών. Παρακαλώ να σεβαστείτε αυτήν την προθεσμία Μπορούμε να ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτηση του θέματος και μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Όπως ξέρετε έχουμε δύο εκθέσεις, δύο σχέδια μάλλον έκθεσης να ζητήσω από όλους σας να ελέγξουμε καταρχήν αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Παρακαλώ λοιπόν να βάλετε τις κάρτες στις σχισμές. Δεν φαντάζομαι να έχουμε πολλές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, αλλά καλού κακού ας το ελέγξουμε. Να ψηφίσουμε μία φορά. Ψηφίζουμε. Ναι. Περιμένω όλοι να βρείτε τις κάρτες σας και να τις βάλετε στις σχισμές. Ε, βλέπω πως κάποιοι συνάδελφοι ακόμα ψάχνουν ε, μέσα στις συλλογές από κάρτες που έχουν. We just... So can we just open the vote and... Vote is open. Vote is open. Ψηφίζουμε. Δεν έχω την κάρτα μου μαζί. Ωραία, λοιπόν, θα βρούμε μια λύση. Ε, μπορείτε να ψηφίσετε διανοτάσιο του χειρό αν δεν έχετε την κάρτα σας. Ωραία, τέλος ψηφοφορίας. Ωραία, λειτουργεί ωραία το σύστημα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Κυρίλοφ. Υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε όπω βλέπετε. Η, τροπολο... η Επιτροπή Προπολογισμού έχει υποβάλει τροπολογίες. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν, να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την έκθεση Κυρίλλου. τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ 7 αποχές εγκρίνεται 9. Ε, τροπολογία 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 από την αποτροπή απασχόληση, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 κατά πίπτη, συγγνώμη δεν το είπα, 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε εδώ τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες, οπότε ε, ψηφίζουμε για την 12 και την budget 5. Υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε. Μία εγκρίνθηκε, εγκρίθηκε. Ωραία. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 12, όπου έχουμε τρεις Ταυτόσιμες τροπολογίε 12, ε, budget 5 και η απασχόληση 12. Ψηφίζουμε υπέρ. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 5 κατά. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αμφιβολίες. Φανέστε Λερόι το ζήτησε. Ωραία, λοιπόν. 13 αγαπητοί συνάδελφοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμός 6 υπέρ καταπίπτει μάλιστα επασχόληση 13 καταπέφτει πάμε στα 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται budget 7 προϋπολογισμός 7 έχει καταπέσει. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 καταπίπτει ή 16 που είναι ταυτόσιμη με την 8 της Επιτροπής Προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της απασχόλησης καταπίπτει, 17 που είναι ταυτόσιμη με την 9 της Επιτροπής Προπολογισμού ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται και προχωράμε έτσι στη 18 γιατί η 15 της επασχόλησης καταπίπτει 18 που είναι ταυτόσιμη με την 10 ε, της προπολογισμού και 16 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ε, επασχόληση 17 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συγγνώμη απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. Εκτιμώντας 1, απασχόληση 1 υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεύτερο εδάφιο, απασχόληση 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας 6, απασχόληση 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 9, ε, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας 11, που είναι ταυτόσιμο με την 2, την ε, προπολογισμό 4, υποσχόληση 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Εκτιμώντας 11, απασχόληση 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Πάμε στην, στο ε, εκτιμώντας 11β, ε, απασχόληση 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκτιμώντας 12, ε, όπου έχουμε την τροπολογία 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και έχουμε την τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Απασχόληση 7 καταπίπτει. Περνάμε στην, το εκτιμώντας 14α, ε, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε η απασχόληση 8 καταπίπτει. Πάμε στο εκτιμώντας 20α, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στις τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμού, στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, περνάμε στον πρώτη τροπολογία υπέρ κατά <coughs> αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προπολογισμό 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τελική ψήφο για το σχέδιο έκθεσης. Οπότε ξεκινά η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 36 ψήφισαν, 41 ψήφισαν, 36 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. So we now move to... Τώρα προχωράμε στο σχέδιο γνωμοδότησης του Γιάννα Όλμπριχτ Λοιπόν, ξεκινάμε με την ε, πρώτη τροπολογία, μάλλον με τη δεύτερη. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Καταπίπτει. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, παράγραφος 4, τροπολογία 4 αποσύρεται, η 5 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 αποσύρεται, πρώτη προφορική τροπολογία Πίπερ. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι είναι σαφής. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε στην παράγραφο 7, αποσύρεται τροπολογία 7, από τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ. Ας ελέγξουμε ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 8, ξεκινά. Λίγη. 7 υπέρ, 33 κατά, άρα απορρίπτεται, αλλά καλό είναι να ελέγχουμε κατά καιρού. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 11, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προχωράμε τώρα στην 2 ε, ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα έχουμε να ψηφίσουμε ολόκληρο το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Λίγη τώρα. 38 υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές, οπότε υπερψηφίζεται και εγκρίνεται το σχέδιο της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία αυτή και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο σημείο 13. δηλαδή τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και ε, προσθέτουμε ε, μέχρι το 2020 τη έκθεση Ρικάρντο Κωστές Λάστρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν. Παρακαλώ να το πράξουν σιωπηλά για να ξεκινήσει η συζήτηση της εκθέσεως. Ρικάντο. Και ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων για τη συνδρομή τους. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría agradecer... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία των ομάδων, τους εισηγητές, τους χιώδης εισηγητές και τις ε, εμπλεκόμενες ε, γενικές διευθύνσεις, στην ΟΚΕ, ε, για την συμβολή τους. Όταν ξεκίνησα την κατάρτιση αυτής της εκθέσεως, συνάντησα διαφόρους, με συγχωρείτε Ρικάρδο, λέει η πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι έχει πολλή φασαρία και είναι πολύ δύσκολο για όποιον είτε μιλά σαν τον εισηγητή είτε θέλει να ακούσει. Ε, έγιναν συζητήσεις με διάφορες ενώσεις, με την Επιτροπή Περιφερειών ε, και με τις απόμακρες ε, ε, παραθαλάσσιες περιοχές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και Απασχόλησης και λήφθησαν υπόψη τα διάφορα θέματα σε αυτή την έκθεση κατά τρόπον ώστε να βρεθεί ε, σημείο συνενέσεως για να καταρτιστεί η έκθεση αυτή για το 2020 ε, αποφασίσαμε στη συνέχεια να προσθέσουμε ε, μια διάσταση που να φέρεται στην πολιτική συνοχή για την επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων του 2020 υπάρχει μία σταθερή ε, πολιτική και μία πολιτική η οποία παρακολουθούνται ε, και εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και αυτή είναι η στρατηγική του 2020 όπου στην αρχή εξετάζουμε την ε, πολιτική και κατακρίνουμε την απουσία αξιολογήσεως των πραγματικών δαπανών την, ε, τονίζουμε την ε, μη αποτελεσματικότητα του προγράμματος και περιμένουμε την ε, έκθεση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να υπάρξει μία αξιολόγηση της επιπτώσεως. Επίσης δεν υπάρχει συμμετοχή των περιφερειακών αρχών και των τοπικών αρχών που δεν έχουν εμπλακεί επαρκώς και η έλλειψη των, της συμμετοχής τους διακινδυνεύει την εφαρμογή της στρατηγικής Λισαβόνας. Τέλος, αναφερόμαστε εις ε, την στρατηγική του 2020 και τις επιπτώσεις και τις, ε, ε, τους συνδυασμούς που είναι τα βασικά σημεία της στρατηγικής για το 2020 και το εχέγγυο επιτυχίας αυτής της στρατηγικής Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να εξετάσουμε τα, όλα αυτά τα στοιχεία γενικά για να μην υπάρχει αποσύνδεση από αυτές τις πολιτικές. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων ζητούμε να αυξηθεί η περιφερειακή και τοπική διάσταση, να προωθηθεί η έρευνα και η παιδεία και να μπορέσουμε να επιτύχουμε το τρίγωνο της γνώσεως και να αποδεσμεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τον βασικό παράγοντα και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όπου χρειάζεται ευελιξία για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε ε, την ε, ε, ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των ε, στρατηγικών προγραμμάτων αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και των διαρθρωτικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο ιδίως τα θέματα που αναφέρονται στη στρατηγική μας διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά αλλά για να διευκολύνουμε, ε, διευκολύνουμε την εργασία της τράπεζας αυτής θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και θα ήθελα τώρα να ακούσω τα σχόλιά σας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το έγγραφό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και προτού ζητήσω από τον Dirk Άνερ που είναι Γενικός Διευθυντής για την Περιφερειακή Πολιτική να λάβει το λόγο θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε ζητήσει από τη διάσκεψη των Προέδρων να αλλάξουν ε, την επικεφαλίδα της εκθέσεως και να προσθέσουν τους στόχους του 2020. Για όσους λοιπόν ε, δεν υπήρχαν εδώ εχθές έχουμε λάβει μία θετική αξιολόγηση από τους ε, Προέδρους των Επιτροπών και τώρα έχει προωθηθεί το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων που αν ε, θυμάμαι καλά θα συνέλθει στις 12 Απριλίου αλλά όποια και να είναι η απόφαση θα υποβάλουμε την έκθεση αυτή για την κατάρτιση στρατηγικής για το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τώρα τον Άννη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο εξέσεως διότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμος ότι έχετε επεκτείνει την έκθεση αυτή για να περιλάβει την Ευρώπη, ε, τη στρατηγική της ε, Ευρώπης του 2020 και εντυπωσιάστηκα από το περιεχόμενο της έκθεσης η οποία ιδίως τονίζει ένα θέμα ότι δηλαδή η πολιτική συνοχή δεν είναι μόνο η πηγή σταθερών επιδοτήσεων αλλά προωθεί την πραγματική συνεργασία που θα προωθήσει την στρατηγική. Επίσης από δικιά μας άποψη το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως άλλωστε και το σχετικό μήνυμα. Ε, στις επόμενες εβδομάδες κυρία Πρόεδρε θα δώσουμε στο Κοινοβούλιο την πρώτη έκθεση προόδου η οποία αναφέρεται στα σχόλια όλων των κρατών μελών για την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος πράγμα το οποίο είναι μια καινοτομία αυτή την ε, περίοδο και οι εκθέσεις μας έχουν δώσει πολλές ε, σημαντικές ε, ε, πληροφορίες σχετικά με το ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα διότι υπάρχουν 230 εκατομμύρια τα οποία έχουν αφιερωθεί στην στρατηγική αντιδράσεως και εις τον προβληματισμό του ποιοι πρέπει να είναι ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ε, στρατηγικής Λισαβόνας για το 2020 διότι μεταξύ των προγραμμάτων των κρατών μελών και των ε, τεκτενωμένων ε, επιτόπου διαπιστώσαμε τα εξής. Θα περιγράψω σε λίγα λόγια για να έχετε ε, συνεκτικές πληροφορίες. Δηλαδή το πρώτο που με ανησυχεί καταρχήν είναι ότι γενικά η εφαρμογή επιτόπου μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ αργή. Και αυτό ο άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Υπάρχουν βέβαια διαφορές μεταξύ των κρατών και αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα από την έκθεση αυτή. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της Λισαβόνας, προχωρούν καλά και μάλιστα σχετικά καλύτερα από το μέσο όρο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παρόλο, παρόλη την κρίση αυτό που ήταν σημαντικό ε, για μας φαίνεται να λειτουργεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μέχρι στιγμής. Και πάλι βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο όπου ε, έχουμε περίπου 27% των ε, αναγκαίων χρημάτων για όλη την περίοδο που έχουν ανατεθεί στα διάφορα προγράμματα επιτόπου, δηλαδή τα χρήματα έχουν δεσμευθεί ε, για τα προγράμματα αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί υποχρεωτικά ακόμη. Αν δείτε λοιπόν ποιο είναι το ποσοστό αφομοιώσεως βλέπετε ότι είμαστε στο 14% το οποίο συγκρίνεται αν μπορεί κανείς να κάνει μία σύγκριση με 20-21% ε, σε σχέση με την περίοδο του 2000-2006, δηλαδή μετά από τρία χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να επιταχύνουμε στα επόμενα χρόνια και θα χρειαστεί ε, εκ μέρους μας μία μεγάλη προσπάθεια, πράγμα το οποίο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ε, για να ανταποκριθούμε στις χώρες που έχουν προβλήματα αφομοιώσεις. Εάν μου επιτρέπετε όμως κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ και να σας, ρωτήσω, να σας ζητήσω και τη δικιά σας βοήθεια κατά τρόπον ώστε το μήνυμα να περάσει και στις χώρες σας και θα ήμουν απανευτυχής εάν θέλετε εάν επιθυμείτε πιο ο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις διάφορες χώρες ε, εγώ και οι συνάδελφοί μου να σας ενημερώσουμε συγκεκριμένα για την κάθε χώρα σας για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά διότι όταν θα γίνει η δημοσιονομική αναθεώρηση και στο το μελλοντικό ο δημοσιονομικό πλαίσιο του χρόνου θα πρέπει όλοι ε, να εξετάσουμε εξετάσουν και το ποσοστό αφομοιώσεως των πόρων που έχουν διατεθεί μέχρι τούδε. Όσον αφορά τη στρατηγική έκθεση, η οποία θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή τέλος Μαρτίου, θα πρέπει να την παρουσιάσουμε πιο λεπτομερώς σε εσά και ε, για μας ήταν μια πλούσια πηγή πληροφοριών και θα ήθελα τώρα να πω ορισμένα πράγματα για τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020 και ε, ουσιαστικά θα ήθελα να σας πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο σχέδιο της εκθέσεως τι πρέπει να γίνει σχετικά με την Ευρώπη του 2020. Όπως είπα ήδη, ε, πιστεύουμε ότι η τρέχουσα πολιτική η οποία έχει καταρτιστεί μαζί με ε, τα σημεία τα οποία έχουν ε, υπογραμμιστεί για τη στρατηγική της Λισαβόνας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020 και θεωρούμε ότι είναι καθήκον της πολιτικής μας να προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε την πολιτική αυτή σε εξελίξεις επιτόπου. Και εδώ αυτή η πολιτική είναι ιδεώδης διότι μπορούμε να πούμε ότι είναι η πολιτική της κοινότητας η οποία μπορεί να περιλάβει διάφορες τομιακές πολιτικές ε, και να τις εφαρμόσει επί τόπου λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της περιοχής και ε, να καταρτήσει συγκεκριμένα προγράμματα. Μην ξεχνάτε ότι η πολιτική συνοχής θα παίξει ένα σημαντικό σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη του 2020 και τη σχετική ατζέντα διότι εφέτος θα έχουμε ε, δύο ανακοινώσεις που θα αναφέρονται σε την ε, ατζέντα της Λισαβόνας καταρχήν όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε μία νέα ανακοίνωση θα κοιτάξουμε συγκεκριμένα πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε τη στρατηγική αυτή σε πρακτικά θέματα επιτρόπου, επιτόπου. Πράγμα το οποίο θα γίνει και με την ε, καινοτομία γιατί είναι ένα από τα βασικά θέματα για την ε, ε, ατζέντα του 2020. Πιστεύω ότι η ε, συνολική εφαρμογή του 2020 ε, η έξυπνη ανάπτυξη, η αηφόρα ανάπτυξη είναι θέματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Γι' αυτό και σκοπεύουμε εδώ να παίξουμε έναν πολύ ενεργό ρόλο. Προς το τέλος του χρόνου, όπως ξέρετε, θα διατυπώσουμε την έκθεση συνοχής μας, όπου έχουμε επίσης στο, σαν στόχο να περιλάβουμε απόψεις που να αναφέρονται εις ε, τις ε, ε, ε, στους προσανατολισμούς μας για το μέλλον και θα τους συνδέσουμε με, με ε, την ατζέντα για το 2020. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω το βασικό ρόλο τον οποίο ε, ε, διαβλέπουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας στη διαδικασία αυτή, όχι μόνο όσον αφορά τις ικανότητές σας σαν συνομοθέτες, αλλά σαν μια κινητήριο δύναμη για να κινητοποιήσει και τους ε, πολίτες και τα κοινοβούλια μας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική έκθεση για να καταρτήσουμε από κοινού έναν απολογισμό για το πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα να σας ενημερώνω τακτικά και κατά τα επόμενα έτη, ίσως δύο φορές το χρόνο, να κάνουμε μία έκθεση σχετικά με το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αφομοίωση της πολιτικής, ιδίως επιτόπου στις χώρες αυτές, διότι αυτό θα είναι ένα από τα βασικά μας θέματα, μία βασική πρόκληση γιατί θα πρέπει να ανταποκριθούμε στους στόχους στους οποίους έχουμε καταρτήσει και να παρουσιάσουμε μία πολιτική η οποία θα μπορέσει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου. Εκ προημίου λοιπόν σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας και για την βοήθεια την οποία ήδη μας έχετε προσφέρει κατά τους τελευταίους μήνες εάν κοιτάξω αυτή τη νέα πολιτική διαπιστώνω ότι στα πλαίσια της Ευρώπης του 2020 ε, βλέπουμε ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να είναι μια πολύ σύγχρονη πολιτική ανάπτυξης. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για το όσα μας είπατε και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο αυτό που μας είπε ο κύριος Γενικός συνάδελφε σε σχέση με τις πληροφορίες μπορείτε να, να βρείτε για το μέρος προελευσής σε σχέση με την ε, πολιτική της συνοχής. Είναι στη διάθεσή σας ο κύριος Γενικός από ό,τι κατάλαβα, πόσο μας είπε επίσης. Κύριε ε, Γενικέ, εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικός ο ρόλος μας έχει ανατεθεί ε, για το όραμα της Ευρώπης του 2020 γιατί τώρα έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και σε σχέση με την εποπτεία της όλης διαδικασίας όχι μόνο με την ε, κινητοποίηση, την προώθηση του, του οράματος αυτού, αλλά ε, νομίζω ότι με την ε, συνεργασία μαζί σας τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο θετικά. Τώρα, θέλω να απευθυνθώ εις τους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτη, κυρία Κοβάλσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αρχίσω. Πρόεδρε, με ευχαριστίες προς όσους συνέταξαν αυτή την αξιόλογη έκθεση. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Ρίξτε μια ματιά στις τροπολογίες μου και θα διαπιστώσετε ότι προσπαθούμε να περιλάβουμε εκεί πάνω από μία απόψεις. Διαπιστώνεται επίσης ότι μειώνονται οι τροπολογίες όσο περνάει ο χρόνος και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Ρίξτε μια ματιά στη συνέπειες της θετικής της Λισαβόνας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αυτό αφορά και την πολιτική για το 2020. γιατί ακριβώς αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος σαν Επιτροπής. Νομίζω όμως ότι σε σχέση με την πολιτική το 2020 δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία, η απαραίτητη προσοχή στην περιφερειακή πολιτική, στις περιφέρειες της Ευρώπης. Άρα θα πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο η υπόθεση των περιφερειών, η διάσταση τη πολιτική του 2020. Κάτι άλλο. Προσοχή να μην ε, εστιάζουν, να μην διαμορφώνουν την πολιτική αυτή με γνώμονα τις πλουσιότερες περιφέρειες. Όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιφέρειες, ακόμα και αυτές που είναι ουραγοί στην, στην ε, ανάπτυξη. Οι πιο φτωχές. Άρα χρειάζεται να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτική το 2020. Τώρα, για να δούμε τους αναπτυξιακούς μας ε, στόχους, χωρίς να ξεχνούμε ότι επιβάλλεται να μην παραμεληθεί ούτε η πολιτική ενέργεια, ούτε η πολιτική μεταφορών, ούτε η πληροφορική. Θα πρέπει να κινηθούμε προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, και να μην ξεχνούμε ποτέ το ευρύτερο τοπίο, την ευρύτερη εικόνα. Η έκθεση επίση μιλάει για την πολιτική της συνοχής και θεωρεί ότι είναι αυτό που πρέπει να πρετανεύσει σαν πολιτική. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε πολλά επίπεδα ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φάσμα είναι πολύ ευρύ. Και είναι πιο μεγάλες τώρα οι διαφορές πρέπει να γεφυρώσουμε από ό,τι στο παρελθόν, γιατί έγινε η διεύρυνση. Αυξήθηκαν, άνοιξε, άνοιξε η ψαλίδα όσον αφορά την ανάπτυξη. Άνοιξε η ψαλίδα μεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό σας λέω ότι και αυτό θα πρέπει να ακουστεί και να υποθεί μέσα από το έγγραφο που εξεργαζόμαστε και έτσι το έγγραφο αυτό να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να τονίσουμε τις προτάσεις μας και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την πράσινη οικονομία. Και το ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της κοινωνίας της γνώσης. Η πράσινη οικονομία φυσικά κοστίζει. Αλλά όπως προείπα, η πολιτική της συνοχής δεν είναι μια ιδέα, ένα ιδεολόγημα αφηρημένο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητείται σε συγκεκριμένη βάση και να καθοριστούν προτεραιότητες και αντίστοιχα η προοικοδότηση. Φυσικά και το προγραμματισμό δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχιστεί η κουβέντα για την έκθεσή μα. Οπότε θα επεξεργαστώ και εγώ το αντίστοιχο στις τροπολογίες για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. επομενο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγώ με τη σειρά μου θα τονίσω ότι ακριβώς όπως είπε και ο εισηγητής από τη φάση 2000-2006 ξεκίνησε μια πολιτική συνοχής που όλο ένα και πιο σημαντική γινότανε. Έχουμε τώρα σαν προτεραιότητα την πολιτική αυτή λόγω της συνέχισης Λισαβόνας, επομένως πάμε για σημαντικές επενδύσεις σε καινοτομία και έρευνα. Έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη οικονομική με ρυθμούς. Πάντως θα πρέπει να έχουμε άμεσες και βιώσιμες λύσεις μια που περνάμε κρίση και έτσι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Επίσης θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να έχουν τέτοια κατάρτιση και εκπαίδευση που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Και το τονίζει αυτό το έγγραφο. Λέει επομένω ότι θα πρέπει να ζητηθεί με ποιο τρόπο οι περιφερειακές αρχές πρόκειται να εμπλακούν στην υλοποίηση της στρατηγικής για το 2020. Εμείς επανειλημμένα τα έχουμε πει. Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από το αν θα γίνει εφαρμογή της σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να ενέχονται και οι περιφερειακές αρχές. Να έχουν και αυτές αρμοδιότητες και ευθύνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από την πολιτική της σύνοχης και από τη στρατηγική του 2020. Έτσι θα πρέπει να εφαρμοστεί στα 2020. Με τα κριτήρια και το πνεύμα της πολιτικής της συνοχής. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση του κύριου Λάστρα. Είναι μια αφετηρία για τον προβληματισμό μας. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Η κυρία Σουέντερ δεν είναι εδώ και άρα έχει το λόγο για Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω είναι σημαντική αυτή η έκθεση που εξετάζουμε. Ε, πρέπει να πάρθουν υπόψη οι εξελίξεις ε, όλο αυτό το χρονικό ε, διάστημα. Ε, το ουσιαστικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι όμως ότι ε, έχουν διευρυνθεί η, η ψαλίδα, η απόκληση μεταξύ των διάφορων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου σημειώθηκε και από μία ομιλήτρια πριν από μένα. Εάν η έκθεση δεν καταφέρει να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί συνέβηκε ε, αυτή η διαδικασία, η οποία είναι υπαρκτή. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Είναι ε, μια υπαρκτή κατάσταση τότε η οποιαδήποτε δουλειά γίνει ε, δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει στο να εκπληρωθούν οι στόχοι της συνοχής που αυτό είναι και ο δηλωμένος στόχος ε, της ε, δουλειάς ε, που κάνουμε. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα πόσο τα ταμεία συνοχής μπορέσαν ή μπορούν να οδηγήσουν σε μια εξισορρόπηση του επίπεδου ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το κριτήριο εκείνο που μπορεί να μας δώσει χειροπιαστά ε, αποτελέσματα για το ζήτημα αυτό και στη βάση αυτή φυσικά να οικοδομήσει κανείς ε, μια προοπτική για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Äh, äh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λέει κυρία Κρέλ. Και εγώ με τη σειρά μου ε, συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη η έκθεσή του και βέβαια θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε το πόσο δύσκολε συνθήκε είναι αυτέ που περιβάλλουν το έργο του. Ε, γιατί είχαμε αυτή την έκθεση δύο πρωτοβουλία και αυτό που θέλαμε ήταν να κάτσουμε και να αναλύσουμε το τι γίνεται με την πολιτική τη συνοχή. Πόσο βοήθησε ε, για την συνθήκη της Λισαβόνας, μια που πολλοί ισχυρίζονται ότι η στατική της Λισαβόνας απέτυχε, χρεοκόπησε δεν πέτυχε τους ε, στόχους που είχαν τεθεί. Και εμείς θέλουμε να γίνει μια δημόσια κρόαση στην ε, Επιτροπή μας, να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα, να τεθεί επί τραπέζι και να συζητήσουμε τα πράγματα. Όμως δεν είχαμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας και έτσι δεν έγινε ποτέ αυτό. Εγώ έχω να σας πω ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτό που θέλουμε, ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια ανάλυση. Μας βόηθησε η στρατηγική τη Λισαβόνα. Τι έγινε, πού, πού, πού φτάσαμε, τι κάνουμε τώρα. Να δούμε τι προτάσει έχει κατεβάσει η Επιτροπή και τι έχει να πει το Κοινοβούλιο. Ότι χρειάζεται δηλαδή μια στρατηγική. Να δούμε τι δεν ολοκληρώθηκε, τι δεν αναλύθηκε, τι πετύχαμε, γιατί ξεκινάμε μια περίοδο νέας δεκαετίας που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε. Ε, εκεί είναι η δυσκολία και γι' αυτό και έχω να απευθύνω συγχαρητήρια προς τον Ρικάρντο γιατί αυτή η έκθεση έχει κάποια άριστα στοιχεία όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να, να διαμορφώσουμε την πολιτική συνοχή από τη μια μέρα στην άλλη έτσι με ένα νομοθέτημα στο γόνατο. Άρα, τι θα κάνουμε, πώς θα ξέρουμε τι πετύχαμε από τους στόχους μας, δεν θα πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα από την αρχή. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πει και ο Ρικάρντο. Πρέπει να έχουμε τις ε, απαραίτητες πληροφορίες και άρα θα πρέπει όλα αυτά εντατικά να τα κοβιδιάσουμε στους αμέσως επόμενους μήνες. Και έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε αλλιώ. ο κόσμος τι θα πει. Θα πει ότι δεν κάναμε αρκετά. Ότι δεν υπηρετήσαμε την πολιτική της συνοχής. Γιατί θέλουμε για όλη την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μια πολιτική συνοχή, όχι μόνο για τι περιφέρειε. Αυτή είναι σωστή προσέγγιση και αυτή είναι οθετή η έκθεση και θα πρέπει μέσα να κάνουμε αυτή την ανάλυση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Χιούμπνερ, με την ευκαιρία που μου δώσατε, κυρία Κρέλ, θα σα πω και εγώ δύο λόγια μετά. Όπω έλεγε ο κύριο Γενικό, Τέλο του μηνό πρόκειται να ολοκληρώσετε αυτή την στρατηγική έκθεση και έτσι θα έχουμε κάποια στοιχεία να τα συγκρίνουμε με όσα έχουμε μέχρι σήμερα. Επίση έχουμε και αυτή την πολιτική έκθεση του Ρικάρντο Κορτέ Λάστρα. Μπα και γίνεται στην επόμενη μα συνάντηση να έχουμε εδώ πέρα ε, τον ε, αρμόδιο επίτροπο και να κάτσουμε να συζητήσουμε με τη βάση τη στρατηγική έκθεση που θα περάσει και από το Συμβούλιο, από ό,τι ξέρω και στην επόμενη συνάντηση κορυφής. Λάμπερτ Φανίστελο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με αυτή την έκθεση, με το περιεχόμενό της και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Αλλά δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος για το πώς γίνεται η συζήτηση. Είμαστε στην Επιτροπή συζητάμε τη Λισαβόνα και την Νέα Στρατηγική 2020, αλλά όπως είπα και χτες στο Συμβούλιο, το παρουσιάζει ως κάτι το οποίο ανήκει στο Συμβούλιο. Δεν το σκέφτονται. Λένε εμπρός. Δέκα χρόνια. Όθηση για δέκα χρόνια. Μα είναι απίστευτο και απαράδεκτο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κρέιλ που είναι η συντονίστρια των σοσιαλιστών. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια βήματα και απλώ να τα δεχόμαστε εμεί. Ίσως λοιπόν θα κάνω μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα να δω τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει από κοινού και έχουν λειτουργήσει σωστά. Ας πούμε, έχουμε κάνει μια παρακολούθηση της εφαρμογής της Λισαβόνας. Εκείνοι παράβλεψαν ε, ότι το 70% των επενδύσεων είναι στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και τους ε, στόχους της Λισαβόνας. Γιατί λοιπόν να μην ε, ακολουθήσουμε την ιδέα που έχει αναφερθεί ότι αν, όπως έγινε και είχαμε και την έκθεση ΚΟΚ που έλεγε τα κράτη Κανένα δεν ήταν υπεύθυνο τότε. Εντάξει, τώρα είναι τα κράτη υπεύθυνα. Και μετά τι έγινε, τα κράτη έκαναν τις ε, διετήσεις εκθέσεις ε, και είπαν ωραία, τα στέλνουμε αυτά στι Βρυξέλλε και χαίρεται και αντίο. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε εμεί μια καινοτομία εδώ πέρα που την έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Γιατί η Ευρώπη να μην κάνει μια συμφωνία με τι περιφέρειες και τις πόλεις ώστε να κάνουν τις προτάσεις για το 2020, να δουν πώς, πώς θα ενεργήσουν πραγματικά. Οι πραγματικοί φορείς πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα ενεργήσουν. Γιατί ποιος είναι υπεύθυνο, όλοι και κανείς. Περιφέρειες, πόλεις κτλ. Ποιος έκανε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης κάθονται εκεί πέρα οι, κάποιοι υπουργοί, κάποιο μέλο τη κυβέρνηση και κάποιε φορέ ούτε καν έρχονται σε επαφή με τι περιφέρειε και τα στέλνουν στι Βρυξέλλε και χαίρονται και αντί όπω είπα και πριν. Είναι πραγματικά αποτυχημένο το σύστημα αυτό. Χαρεοκοπημένο και αποτυχημένο. Θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική περιφερειακή που να φτάσει μέχρι το 2020, ναι, να την κάνουμε. Εγώ δεν είμαι κατά το, να βάλουμε και τα χρήματα για αυτά να τα προβλέψουμε. Δεν είμαι κατά να έχουμε μια πολύ πολυεπίπεδη προσέγγιση όπου τα, κράτη και οι περιφέρειες θα λαμβάνουν μέρος στη δράση και αν κάποια περιφέρεια ή κάποια κράτη πούνε ναι εντάξει εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στη δράση, γούστα τους και καπέλο τους. Δική τους είναι η επιλογή. να κάνουμε μια δράση όπου οι εταίροι πραγματικά θα επενδύουν και θα το θέλουν. Όχι θα κάθονται όλοι ήσυχα και ξαφνικά θα έχουμε απλώς μια χοροδία δηλαδή όπου κανείς δεν τραγουδά αλλά υπάρχει ε, ε, ε, δεν θέλουμε να είναι αυτό η Ευρώπη Εγώ θέλω λοιπόν μια συνεργασία με τις περιφέρειες και τις πόλεις, μια Ευρώπη όπου θα συμβάλλει για να βγούμε από αυτή τη συζήτηση όπου όλοι στριφογυρνάμε γύρω από το θέμα, αλλά κανένας δεν αποφασίζει. Να έχουμε μια-δύο παραγράφους. Εγώ θέλω λοιπόν περισσότερη ορατότητα. Όπως λένε και οι Γερμανοί, Δηλαδή να είμαστε κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό και θα κάνω κάποιες τροπολογίες όπου θα λέει ναι, η περιφερειακή πολιτική έχει κάποιες ιδέες και ίσως και ο κύριος Άρμπνε στην συζήτηση για τη αναθεώρηση, την οικονομική αναθεώρηση. Με το πολύ πολύ κακό αυτό έγγραφο που είχαμε, που ήταν τρελό εκείνο το έγγραφο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, το είπα τώρα, τελείωσε. Εμείς ευχαριστούμε Λαμπέρ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Φανίθελτο, γιατί θεωρώ ότι αν κανείς ε, ε, μελετήσει την στρατηγική της Λισαβόνας, θα συμφωνήσει ότι υπάρχει εδώ ένα έλλειμμα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα έμπνευσε. Δεν υπάρχει κίνητρο. Οπότε, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, ότι το Κοινοβουλίο θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική του 2020, ακριβώς όπως και το Συμβούλιο. Επίσης ώρες, ισότιμα. Η στρατηγική αυτή θα πετύχει μόνο εάν δεν περιοριστεί η υπόθεση σε, σε, σε παιχνίδι κοινοβουλίου και συμβουλίου, αλλά αν εμπλακεί και ο λαός της Ευρώπης. Επομένως, ε, θα πρέπει και εμείς, σαν Επιτροπή Περιφερειακή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό και εγώ σας συνιστώ να εξασφαλιστεί ότι ο παράγων περιφέρειας να παίξει ένα ρόλο κλειδί στη στρατηγική του 2020. Κύριε Γενική, τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αυτή η έκθεση ήταν αναλυτική. Θα πρέπει επίσης να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα από κάποια παλιότερα περιφερειακά προγράμματα. Χρειαζόμαστε όλα τα δεδομένα πληροφορίε που υπάρχουν και ελπίζω να μου απαντήσετε σε αυτό που θα να μάθω για στρατηγική του 2020. Ό,τι δηλαδή. Εάν κάτσουμε και δούμε τι προγράμματα ισχύουν και τρέχουν σήμερα. Μήπως τα προγράμματα που τρέχουν σήμερα δεν λαμβάνουν υπόψη τις ε, περιφερειακές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα αναδεχθεί η καινούργια πολιτική το πνεύμα της προτεραιότητας της προηγούμενης πολιτικής. Να δούμε μόνο τι θα γίνει κατά το πρώτο ένα τρίτο της καινούργιας ε, στατικής για το 2020 να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει κάποια συνέχεια και προσαρμογή των προηγουμένως ισχυσάντων. Γιάν Άλμπριχτ και κατόπιν Ιωάκιμ Τσέλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου εγώ να πω κάτι λίγο προκλητικό. Δηλαδή, ακόμα τον κόσμο να λέει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε. Ξέρετε, αποτυχημένη τη θεώρησε ακόμα και ο πρώτος Μπαρόσο. Γι' αυτό και σας λέω ότι αν πρόκειται να συνδεθεί η στατική της Λισαβόνας με την πολιτική της συνοχής, τότε θα πρέπει εδώ να μην τα ανακατεύουμε όλα και να χρησιμοποιήσουμε χωριστά και να μελετήσουμε χωριστά το κάθε τμήμα αυτής της έκθεσης. Γιατί αν κάτσει κανείς και δει το ιστορικό πλαίσιο της στρατηγικής Λισαβόνας, δεν είχε συνδεθεί ανέκαθεν ε, η στρατηγική της Λισαβόνας με την πολιτική της συνογής. Είχαμε την, ε, ανοιχτή, τον ανοιχτό συντονισμό, ε, είχαμε ιδιαίτερος πολλές ευθύνες που έπεφταν στα κράτη-μέλη. Και προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε τις περιφέρειες και τις μεγάλες πόλεις. Και σας παραπέμπω στην έκθεση και στην ε, λεγόμενη μαύρη λίστα. Τώρα να δούμε κατά πόσον θα λισαβονοποιηθεί η καινούργια στρατηγική. Θα πρέπει από την αρχή να πάρουμε σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να χτίσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές με κάποια θεμέλια γερά. Αλλιώς δεν θα βγει τίποτα. Συντονισμός, πόροι, κοινά μέσα πολιτικής. Είχαμε τα δεσμευμένα ποσά, με τα παλιά κράτη-μέλη, έτσι δουλεύαμε παλιότερα. Επομένω, τώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, και όπω τα λέει και η κοινωνία χθε, έχουμε βασικά δύο στρατηγικέ. Και ακριβώ τώρα πρέπει να διορθώσουμε το λάθο που κάναμε. Ότι δηλαδή δεν βάλαμε την πολιτική τη συνοχή μέσα στη στρατηγική τη Λισαβόνα. Γιατί νομίζω ότι αν το είχαμε κάνει αυτό θα σωζόταν τροποντινά η στρατηγική τη Λισαβόνα. Άρα τώρα τα δύο αυτά πράγματα έχουν αυτό το, το, το, ένα σύνολο, το ενιαίο, έχει γίνει δύο χωριστά. Προσοχή μας το γιατί διατρέχουμε τον ε, κίνδυνο να καούν τα χλωρά με τα ξερά. Να κάτσουμε τώρα επομένω να δούμε πώς θα αξίζει τη Λισαβόνα, να, ε, την ενημερώσουμε και να δούμε πώς θα κάτσουμε να ξεδιαλέξουμε το ποια αξιόλογα στοιχεία υπήρχαν στην πολιτική της Λισαβόνας και να τα βάλουμε στην στρατηγική του 2020, τουλάχιστον για την πρώτη δεκαετία, γιατί εδώ λέμε για τις περιφέρειες, μας ενδιαφέρουν, αλλά επίσης μιλάμε και για, τις, ε, για το, το, το, αστικό περιβάλλον της πόλης δηλαδή, Ας κάτσουμε λοιπόν να σκεφτούμε ότι έχουμε αυτή τη, τη στρατηγική ό,τι έχει να προσφέρει η Λισαβόνα να το αξιολογήσουμε και ταυτόχρονα να ξεσκαρδάρουμε τα, τα, τα λάθη, τα αρνητικά. Έτσι, αν έχουμε αυτό το διαχωρισμό θα πάμε καλά. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αν προερχόμαστε από κάπου και θέλουμε να πάμε σε ένα καινούριο σημείο πρέπει καταρχήν να αναλύσουμε το παρελθόν και με αυτό ε, είμαι ευγνώμων στον εισηγητή γιατί ακολούθησε αυτή την πρόταση. Εδώ μιλάμε πάρα πολύ για την περιφέρεια και προτού έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχα ασχοληθεί πολιτικά με την περιφέρεια και ε, ήμουν αρκετά δραστήριος για μένα η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν κάτι που διάβαζα στην εφημερίδα. Δεν ήταν δηλαδή ε, μία ε, βάση για την καθημερινή μας πολιτική δράση. Αφενός, αφετέρου, Πιστεύω ότι είναι καθήκον της στρατηγικής να καθορίζει στόχους και εδώ συμφωνώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες. Αν στόχος της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ε, να, ε, αναπτύξει την Ευρώπη σαν το πιο δυναμικό χώρο, ο στόχος αυτός απέτυχε. Ε, βέβαια υπήρξε μια οικονομική ε, κρίση και αυτό δεν μας βοηθά διότι η ίδια κρίση έπληξε ε, και ακόμη περισσότερο άλλους χώρους πέραν του ευρωπαϊκού. Άρα στρατηγικά ποια είναι τώρα η πρότασή μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτούς τους στόχους ε, ή θα αναζητήσουμε νέους διότι ε, θέλουμε να υπάρξει μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της καινοτομίας αλλά γι' αυτό πρέπει να συμπράξουν όλοι εφόλων των επιπέδων ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών και δεν θα το πετύχουμε με το να είναι απλός κοινοτικός στόχος διότι ε, στη Γερμανία Γερμανία και περιφερειακά ο στόχος του 2020 είναι αρνητικός γιατί ε, υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι συνεδριάζουν στη Γερμανία στο, στη Γερουσία ε, που απέπεψαν εχθές νομοθεσία η οποία θέτησε κίνδυνο την αρχή της επικουρικότητος. Εάν λοιπόν ε, ε, ε, υπάρχουν ε, ήδη επιφυλάξεις από μία τόσο ισχυρή, ισχυρή περιφερειακή αρχή και αυτό το έχω διαπιστώσει και στο Bundestag, δηλαδή στη Βουλή στη, Γερμανία, τότε πρέπει να προβληματιστούμε. Και ε, χθες ο αξιότιμος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Ζέρζι Μπούζ, Μπουζέκ ε, αναφέρθηκε εις τους υπουργούς ε, των ε, γερμανικών κρατηδίων και μας είπε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ασχολ... τους ομοσπονδιακούς υπουργούς μάλλον της Γερμανίας και είπε ότι αυτό που πρέπει να μας υποκινήσει πρέπει να είναι στην Ευρώπη ο ανταγωνισμός. Αυτό πρέπει να μας εμπνεύσει. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η πολιτική συνοχή χρειάστηκε να επιλύσει ορισμένα προβλήματα, σαν αυτά που είπε ο κύριος Όλμπριχτ. δηλαδή ε, την ε, αφομοίωση 12 νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τους πόρους που διέθετε το Ταμείο Συνοχής. Τώρα όμως είμαστε 27 και το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε στόχους οι οποίοι να συνδυάζονται με, την με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί είναι καλύτεροι από μας και άρα πώς θα προωθήσουμε την πολιτική συνοχή θα είναι ένα εργαλείο κατανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα πάρουμε ό,τι υπάρχει σε κάποιο σημείο για να μπορέσουμε να, να προσφέρουμε σε ε, περιοχές που δεν υπάρχει ή χρειάζεται ένας πιο μεγάλος στόχος, ένας πιο ολοκληρωμένος στόχος. Ασχέτως δηλαδή που βρίσκονται οι περιφέρειες θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς και αν εκεί επικεντρωθούμε στην καινοτομία, στην πολυμορφία την οποία έχουμε στην Ευρώπη. Αν όλα αυτά μπορούμε να τα προωθήσουμε και να τα αναβαθμίσουμε, αν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση στην Ευρώπη, τότε θα μπορέσουμε να ωφελήσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν τα κατάφεραν τόσο καλά στην πρώτη φάση διότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσουμε ε, στόχους στις περιφέρειες που χρειάζονται ακόμη την ε, βοήθειά μας ε, ώστε να μην εκτίθενται συνέχεια στο διεθνή ανταγωνισμό και για να μπορέσει να υλοποιηθεί πραγματικά η πολιτική συνοχή και αυτή είναι η συζήτηση που πιστεύω πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Ρικάρντο Λάστρα διότι συνέταξε μια προκλητική μια έκθεση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γιατί σας τα λέω αυτά διότι πρώτα πρώτα θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα της στρατηγική της Λισαβόνας. Να κάτσουμε για να ζυγίσουμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της στρατηγικής και να κάτσουμε να δούμε τι μας λείπει ούτως ώστε να προχωρήσουμε προς άλλες επιτυχίες. Λείπει η πολιτική διακυβέρνηση. Αυτό όμως νομίζω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας βελτιώνεται. Επίση, είναι και θέμα κάποια οικονομική διακυβέρνηση και ήρθε ο Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου και μας τα εξήγησε τις προάλλες. Αλλά όμως αυτό δεν ήταν να το να γίνει ε, χωρίς και ενάντια στις περιφέρειες. Χρειάζεται μια στρατηγική η οποία να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να γίνει ένας ε, ουσιαστικός, σημαντικός παίκτη στην παγκόσμια σκακέρα. Ε, αλλά χρειάζεται να υπάρχει κάποια συνοχή και συνέπεια στην ε, διακυβέρνηση την πολιτική να μην έχουμε μόνο τις δηλώσεις προθέσεων, οπότε εάν τελικά η στατική για το 2020 αφαιθεί στο Συμβούλιο χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο, να έχει απλώς το ρόλο του, του να εγκρίνει την πολιτική, τότε δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε ότι στο Συμβούλιο κυριαρχούν οι εθνικές πολιτικές. Εξού και η επιλογή των επιτρόπων, εξού και οι προστριβές των ε, κρατών μελών σε σχέση ας πούμε με την έξοδα από την κρίση. Εθνικές λοιπόν είναι οι λύσεις που δίνει το Συμβούλιο. Άρα έτσι όμως χάνεται η συνέπεια χάνεται το ότι θα πρέπει να προβάλλεται μια στρατηγική ενωσιακή και όχι των κρατών μελών. Συνάδελφε. Μιλούμε με λόγια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όμως Εάν όλα αυτά δεν διατυπωθούν ξεκάθαρα εγγράφως τότε σε σχέση με Κίνα και με ΙΠΑ δεν μετράμε. Είναι αστείε μας επιδόσεις μα όσον αφορά την διακυβέρνηση. Οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί έχουν διακυβέρνηση. Εμείς δεν έχουμε. Για να δούμε επομένως πώς θέλουμε να βγει από την κρίση η Ευρώπη. Δεν θα βγούμε εάν ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Να κάτσουμε και να δούμε τι περιφέρειες θέλουμε για την Ευρώπη. Ποια είναι η ιδεώδης ε, λύση. Όχι, δεν θα μας βοηθήσει όμως η εθνική σύλληψη των πραγμάτων. αυτού του είδου η σύλληψη των πραγμάτων εξυπηρετεί μόνο ορισμένα κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ούτως ώστε να καθοριστεί, να περιχαραγωθεί μια τέτοια στρατηγική για το 2020 και έτσι να μπορούμε να καταληφθούμε την ευκαιρία. Και το 2020 να μην έχουμε να κάτσουμε να κάνουμε υπολογισμό σε μια νέα αποτυχία, Πρόεδρος. Έρικα Μάνερ esittelijälle erinomaisesta työstä ja hyvästä Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά, είναι πάρα πολύ καλή η έκθεσή σας. Αυτές οι ε, παρεμβάσεις ήταν πάρα πολύ αξιόλογες και εγώ επομένως δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα ίδια. Η στρατηγική του 2020 χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία, το έχουμε αυτό επαναλάβει και όσον αφορά την συνθήκη της Λισαβόνας και τη στρατηγική μάλλον της Λισαβόνας, όχι, δεν απέδωσε, δεν λειτουργήσε όπως θα θέλαμε. Γιατί αυτό. Απλώ γιατί τα κράτη-μέλη δεν στρατεύτηκαν όπω θα έπρεπε για αυτή την ε, πολιτική. Τώρα, όσον αφορά την ε, στατική του 2020, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πέσουμε στα ίδια λάθη. Θα πρέπει να τεθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι. Έχουμε ένα σωρό αξιόλογε ε, ιδέε που αναφέρθηκαν, πάρα πολύ αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι. Επίση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του, του, του, του καρότου και του μπαστονιού για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Στην πράξη επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μαστίκι το καρότο και όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τον κοινοτικό. Θα πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες. Θα πρέπει να πάρει προτεραιότητα η στρατηγική του 2020 για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της. Επίση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνέργεια, να εξασφαλίσουμε συνέπεια, συνοχή μεταξύ των διαφορετικών ε, τρόπων χρηματοδότησης και στα πλαίσια της διαρθρωτικής πολιτικής να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να προβλέψουμε πρώτα-πρώτα κάποιες δράσεις της στρατηγικής αυτής. Και να μπορέσουμε βέβαια να κινητοποιήσουμε τις περιφέρειες και τους τρόπους χρηματοδότησης που έχουμε επιτόπου για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριος Βλάσακ, εγώ θέλω να επανέλθω στα πιο βασικά στοιχεία της έκθεσης. Τι έχει πετύχει η πολιτική της σου ούτως ώστε να συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων της πολιτικής της Λισαβόνας. Αυτή η κουβέντα θα πρέπει να γίνει. Πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι ο κύριος Λάστρα σε αυτή τη γραμμή πλεύσης κινήθηκε. Έχουμε πόρους, έχουμε μέσα πολιτικής που επιστατεύτηκαν πρόσφατα πρόσφατα, άρα δεν έχουμε κάποια δεδομένα για να ζυγίσουμε τι έγινε. Εμείς πάντως προσπαθούμε. Ολοκληρωμένη προσέγγιση, εταιρική σχέση, επικουρικότητα, όλα αυτά είναι μεταβλητές που θα πρέπει να συνδυαστούν και να κάτσουμε και να απευθυνθούμε στο κάθε κράτος μέλος χωριστά και να τους και να ρωτήσουμε, να ψάξουμε να βρούμε τι προτεραιότητες έταξαν. Ελήφθησαν υπόψη προτεραιότητες των πόλεων. Υπήρξαν κάποια σχέδια και προγράμματα ολοκληρωμένα. Μήπως κάποιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν καλύτερα από άλλους. Και η αξιοποίηση των πόρων πώς έγινε. Πήγανε σε καλή μεριά οι πόροι που ήταν διαθέσιμοι. Μήπως δήμοι και κοινότητες θα έπρεπε να εμπλακούν περισσότερο στη διαχείριση των, πόρων τους. Νομίζω μόνο το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ το έκαναν αυτό. Γιατί δεν έγινε το ίδιο κι αλλού σε άλλα κρατημέλη. Φοβόντουσαν κάτι και δεν το έκαναν. Τζέρεμι, Τζέσικα. Ε, το θεμέλιο είναι κάποιες ε, πάρα πολύ σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά περιορισμένη χρήση τους. Κι όμως το μέλλον είναι αυτή η κατεύθυνση. Ποιος ήταν ο φραγμός που δεν ε, χρησιμοποίησαμε αυτές τις φρέσκες μοντέρνες ιδέες, κάτι τελευταίο τώρα. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς οι μόνοι που απασχολούν αυτά τα προβλήματα. Και η Επιτροπή των Περιφερειών και οι ΟΚΙ ασχολούνται με τα ίδια προβλήματα. Ας κάτσουμε να ρωτήσουμε και αυτού μας πώς βλέπουν τα πράγματα και μετά να κάνουμε την ανάλυση μας. Το είπε η συνάδελφο που ζήτησε να γίνει η ακρόαση, η μήνυα ακρόαση τέλο πάντων. Είναι πολύ καλή έκθεση. Και επομένως να κάτσουμε να πάρουμε αυτή την έκθεση, να τη χρησιμοποιήσουμε ε, για να αναλύσουμε το θέμα ή να προβούμε σε κάποιες συστάσεις για το πώς θα έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση των κοινωτικών πόρων. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή ιδίω για το σημείο 14 διότι μέχρι στιγμής δεν το αναφέραμε παρκώς όταν μιλάμε για τη στρατηγική του 2020. Εχθές συζητήσαμε για ανταγωνισμό, για αύξηση ε, και ε, δεν είχα ακούσει ποτέ να μιλάμε για τους ανθρώπους. Ε, το θέμα είναι γιατί θέλουμε τους ανθρώπους, γιατί δίνουμε τόση σημασία στον ανταγωνισμό για να μπορούν να υποφεληθούν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην περιφερειακή πολιτική ε, αυτά τα θέματα τα διαβάζουμε απλώς στις εφημερίδες. Θα πρέπει στην περιφέρεια οι άνθρωποι να μπορούν ε, να αντιληφθούν τι μπορούν να αποκομίσουν όλοι από αυτά τα προγράμματα. Είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί. Η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη έχουν σημασία μόνο εάν μπορούν να υποφεληθούν οι άνθρωποι σε όλες τις περιοχές. Γι' αυτό και χρειάζεται ανακατονομή, όχι μόνο περιφερειακά, αλλά ανακατανομή και από εκεί που υπάρχει όφελος, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι συμβάλλουν ή αυτοί που δεν μπορούν να συμβάλλουν λόγω ελλείψεων ή αδυναμιών διότι ορισμένα από αυτά μπορεί να σας φέρονται κάπως ε, απλοϊκά αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους δεν μιλάμε μόνο για τεχνικά μέτρα και βελτίωση διαδικασιών αλλά πρέπει να δούμε τι περισσεύει δηλαδή ε, τι θα επωφεληθεί ο Ευρωπαίος από αυτά τα οποία κάνουμε και γι' αυτό ε, σας ευχαριστώ χωριστό διότι η ανταγωνιστικότητα δεν θα υπήρχε στην Ευρώπη αν δεν σκεφτόμασταν τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάλεμπαχ. Ευχαριστώ κυρία Κάλεμπαχ. Καλό θα ήταν ίσως να ζητήσουμε μία αντίδραση από τον κύριο, που, κύριο Άντνερ. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε γιατί η συζήτηση αυτή ήταν πολύ επικοδομητική για μένα και θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά τα σημαντικά και νομίζω ότι το είπε η κυρία Τρίλ ε, για να δούμε τα γεγονότα, ας τα βάλουμε στο τραπέζι και ας τα αναλύσουμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο θα έχουμε πολλές δυνατότητες διότι τέλη Μαρτίου θα έχουμε τη στρατηγική έκθεση μετά στις 19 Απριλίου ελπίζω ότι θα έχουμε τις εκθέσεις αξιολογήσεως που συγκεντρώνουν όλα τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει σχετικά με την περίοδο 2000-2006 και όπου διαγράφεται η κατάσταση ε, της στρατηγικής Λισαβόνας και περαιτέρω στους ε, στόχους της ε, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολλά θέματα τα οποία τίθενται και τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. νομίζω ότι ο κύριος Όλμπριχτ έκανε το σχετικό σχόλιο και ο κύριος Τσέλερ και ορισμένα άλλα μέλη ε, της Επιτροπής. Είναι ε, ατυχές ότι η πολιτική συνοχής είχε ρητός συνδεθεί με την στρατηγική της Λισαβόνας μόνο για την περίοδο 2006-2013. Μου είχατε πει πολλές φορές κυρία Πρόεδρε όταν επισκεφτόσασταν τις περιφέρειες πόσα λίγο είχε, ήταν ενημερωμένοι όλοι για την στρατηγική, για τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα, για τις συζητήσεις οι οποίες Δηλαδή, υπήρχαν σε σχετικά με την στρατηγική 2007-2013, δηλαδή ε, πώς αυτό έγινε πιο συγκεκριμένο για, ε, ε, για τις περιφέρειες. Και ε, πρέπει η στρατηγική αυτή και οι στόχοι της να διαδοθούν εις ε, τις περιφέρειες από την αρχή. Και αυτό θα είναι ε, το καθήκον της πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Χαίρομαι διότι διαπιστώνω ότι παρόλο που η στρατηγική του 2020 αναφέρεται σε προτεραιότητες και στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, ανταγωνιστικότητας, ε, καινοτομίας κτλ. προχωρά και περαιτέρω. Δηλαδή περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα ε, τις ε, κοινωνικές ζημίες και επίσης περιλαμβάνει σε μία στρατηγική στην ε, ε, διάσταση της περιβαλλοντολογικής ε, αηφορίας. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Κρίμας που η περιφερειακή πολιτική χρειάστηκε τόσο χρόνο για να υιοθετήσει τη στρατηγική της Λισαβόνας. Δέστε τις ημερομηνίες. Ξεκινήσαμε το 2007. Στο τέλος του 2007 υιοθετήθηκαν τα προϊόντα και μετά τα προϊόντα αυτά άρχισαν να εφαρμόζονται ε, και ε, τώρα ε, στο τέλος του 2009 και τώρα μόνο ένα μικρό μέρος από ό,τι διετίθετο στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής έχει χρησιμοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα μπορούμε να ε, ε, να δούμε τη στρατηγική της Λισαβόνας και να την αντικαταστήσουμε με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 χωρίς όμως να είχαμε την δυνατότητα να αναλύσουμε ρητός τη διασύνδεση της στρατηγικής Λισαβόνας και της ε, περιφερειακής στρατηγικής. Βεβαίως η περιοχή συνοχής είναι μια αυτούσια πολιτική και άλλωστε πολλοί είπαν και πολύ σωστά ότι είναι ε, μία έκφραση ε, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη χωρίς όμως να μιλάμε ε, για ελεμοσύνη. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Όταν λοιπόν κοιτάμε τις αξιολογήσεις της περίοδου 2006 μία από τις φράσεις τις οποίες έχω διατηρήσει στο μυαλό μου είναι ότι ακόμη και αν χρηματοδοτήσουμε ή ακόμη και αν η αλληλεγγύη ενισχύεται στις περιοχές όπου είχε μείνει πίσω η εξέλιξη θα πρέπει να υπάρχει κανείς, ε, θα πρέπει να εξετάσει κανείς το σύνολο διότι εφόσον είμαστε σε έναν ολοκληρωμένο κόσμο δεν μπορούμε απλούστατα να βλέπουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να δούμε πόσο θα προσεγγίσουμε τις διάφορες περιοχές προς το μέσο όρο αλλά αυτό που λέγεται στο 2020 είναι ότι θα έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνέχεια όπου υπάρχουν νέες προκλήσεις άρα αυτό που θα πρέπει να εντοπίσουμε στο μέλλον είναι πόσο θα ισοσκελίσουμε τους διάφορους αυτούς στόχους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι και θα πρέπει να ε, επιτευχθούν συγχρόνως. Εάν αυτό το επιτύχουμε τότε είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε πολύ αποτελεσματικά ή στην μελλοντική η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατά πολύ είναι αυτό το οποίο ε, επιζητά η στρατηγική του 2020. Θα πρέπει δηλαδή να αναπτύξουμε την κοινωνία μας, ε, την ε, οικονομία μας περαιτέρω και επανερχόμαστε στους όρους της συνθήκης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ισοσκελισμένα και ισορροπημένα. Εάν λοιπόν προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πετύχουμε τους στόχους αυτούς στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Είμαι αισιόδοξο, κυρία Πρόεδρε και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον εισαγητή για το σχέδιο της εκθέσεώς τους. Πριν να δώσω το λόγο στον επόμενο μελητή, θα ήθελα και εγώ ίδια να πω δύο λόγια και να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, Κύριε Γενική Διευθυντά, αναφέρατε ότι ορισμένοι διαφοροποιούν ανάμεσα στην συνθήκη που λέει ότι θα πρέπει να στοχεύουμε με την περιφερειακή πολιτική και την περιφερειακή πολιτική να περιορίζουμε τις ε, ανισότητες. Αυτό κάνουμε και με την ε, στόχους της Λισαβόνας. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμιά αντίφαση μέσα σε όλα αυτά. Γιατί τι σημαίνει με μείωση των ανισοτήτων. Δηλαδή να αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές γρηγορότερα από τις άλλες. Και σήμερα για να υπάρχει ανάπτυξη με έναν βιώσιμο τρόπο, δηλαδή που θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο και δεν θα χαθεί, ε, απέναντι στην Κίνα ή την Ινδία, πρέπει να επενδύσουμε σε διάφορα πράγματα που επενδύαμε πριν και 20 χρόνια. Δηλαδή, καινοτομίες όσον αφορά την επάρκεια σε ενέργεια και τα πράσινη ενέργεια και ούτω καθεξής. Το κάνουμε αυτό λοιπόν με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά ανταποκρινόμαστε και στις παγκόσμιες προκλήσεις που δεν περιμένουν για μας. Εμείς πάντοτε πρέπει να τις προλαβαίνουμε, όχι σε σχέση με τους γειτόνε μας μόνο. Η Πολωνία είναι γειτονική με την ε, ε, Γερμανία και με την Ουκρανία από την άλλη μεριά, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και με άλλε χώρες που είναι πιο ανταγωνιστικές από εμάς το Δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε τη συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι η αρχή αυτής της συζήτησης του 2020 είναι και η αρχή για τον προϋπολογισμό, η συζήτηση μάλλον για τον προϋπολογισμό. Αυτό που έχουμε εδώ για το 2020 και τα κονδύλια είναι πιθανότατα ο προϋπολογισμός του, της Ένωσης. πρέπει να λυθούν τα προβλήματα στις δημοσιονομικές αγορές. Θα είναι πρόκληση να βρούμε χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Και στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί καλά ο προπολογισμό της Ένωσης. Ποια είναι η επιλογή για το 2020 με βάση αυτό τον προπολογισμό. Ήδη θα το περικόψουμε σε ένα σύνολο τομεακών ταμείων. Θα φτιάξουμε νέα ταμεία και πιθανότατα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρξουν νέε αρμοδιότητε που θα κοστίσουν πολύ και θα είναι και χρονοβόρα πράγματα όλα αυτά και θα πρέπει και να βρούμε και την ομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν για να διοικεί τέτοιο είδους ε, ταμεία, είτε θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους παγιωμένους μηχανισμούς ε, όπως η πολιτική συνοχή στους οποίους επενδύουμε εδώ και χρόνια. που ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια. Είναι μια πολιτική που στη χρηματοδότησή της ξεκινά με στρατηγικούς στόχους. Ε, μετά αυτοί προσαρμόζονται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες και τέλος μέσω των διαπραγματεύσεων βρίσκουμε τον τρόπο για να κατανείμουμε τα χρήματα και έχουμε και τους όρους που είναι εξαιρετικό και δυνατό όπλο. Έχουμε το μηχανισμό για να ελέγξουμε και έχουμε και το μηχανισμό για να βοηθήσουμε. Γιατί η γάμα δέλτα απασχόληση, περιβάλλον, έχει ένα σωρό κόσμο που μπορούν να πάνε επί τόπου και να βοηθήσουν αυτούς που πρέπει να εφαρμόσουν τα προγράμματα. Έχουμε λοιπόν πολιτική, μηχανισμό εφαρμογής πολιτικής. Γιατί λοιπόν να ψάχνουμε και να εφευρίσκουμε νέα πράγματα και να δαπανίσουμε 10 χρόνια για νέα μηχανήματα χάνουμε απλώς χρόνο. Ανοιχτή μέθοδος ε, συντονισμού, ακόμα και με αυτές τις αλλαγές τώρα που έγιναν μετά από το 2005. Και πάλι αποτελεί ένα πολύ ελαφρύ μηχανισμό που δεν πιστεύω ότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. ώστε να ολοκληρώσουμε τους στόχους. Αυτά λοιπόν. Νομίζω αυτή είναι μια πολιτική που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη. Και όπως έλεγε και ο Λάμπερ και άλλοι, είναι μια πολιτική που θα πρέπει να δώσει και την ευκαιρία στη νέα συνθήκη, που είναι η συνθήκη η οποία λέει πως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους πολίτες τώρα. Ε, δηλαδή ε, τους πολίτες, όχι μόνο τοπικές αρχές και εταίροι, αλλά οι πολίτες οι ίδιοι. Ποιοι λοιπόν μπορούν να καταφέρουν την συμμετοχή των πολιτών. Αυτή η πολιτική που είναι παρούσα και επιτόπου. Νομίζω ότι οποιοδήποτε πιστεύει πως μπορούμε να φτάσουμε αυτούς τους στόχους με διαφορετικούς στόχους, απλώς κάνει λάθος. Και θα δώσω το λόγο στον Ρικάρδο, ώστε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βεβαίω και λαμβάνει υπόψη όλε τι ε, απόψει των συναδέλφων. Όλα όσα είπατε στη συνάντηση τη Επιτροπή μα για την έκθεσή μου, γιατί νομίζω ότι επρόκειτο για πάρα πολύ ενδιαφέρον feedback αυτό το οποίο μου δώσατε όσον αφορά την έκθεσή μου και βεβαίω δεν μπορώ να παραλείψω να ευχαριστήσω και την κυρία Φίμπνερ, την πρόεδρό μα, γιατί και αυτή αποφασιστικά και σταθερά με ενθάρρυνε ε, Ευχαριστώ έργο για την Επιτροπή μου επίσης. Πρέπει να σας πω καταρχήν κάποιες παρατηρήσεις μου για αυτά τα οποία μου είπατε. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για κάποια έκθεση που αφορά τη στρατηγική του 2020, αλλά το πώς μπορεί να συμβάλλει η πολιτική της συνοχής σε αυτή την στρατηγική. Υπάρχει εδώ πέρα μια διαφοροποίηση πρέπει να κάνουμε. Και ακριβώ γι' αυτό προσφέρει ενδιαφέρον η συζήτησή μα. Γιατί είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι να τα συζητά και να γίνονται λόγοι περισσότερε τέτοιε συζητήσει γιατί θα πρέπει το νωρίτερο δυνατόν να πάρει το δρόμο τη αυτή η στρατηγική και να προχωρήσουμε σε μια υπόθεση καθόλου εύκολη για όλη την Ευρώπη. Ε, συμφωνούμε για το ρόλο των ε, τοπικών αρχών και των περιφερειών και ότι θα πρέπει να εμπλακούν όλες αυτές οι, οι αρχές και φορείς σε αυτή την τόσο στρατηγική σημασία πολιτική. Ε, κύριε Λαμπέρτ, συμφωνούμε για το ότι θα πρέπει να αγκαλιάσουν οι πολίτες αυτή την πολιτική, την πολιτική της συνοχής που είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Κύριε Άλμπρεχτ, επίση συμφωνώ ότι η πολιτική της συνοχής έσωσε πολλά στοιχεία της πολιτικής της Λισαβόνας και χρειάζεται όμως να γίνει ένα συντονισμό μεταξύ όλων των σχετικών συγγενών πολιτικών γιατί νομίζω ότι το μοναδικό υποχρεωτικό στοιχείο και αναγκαστικό της πολιτικής της της αγώνας ήταν αυτή η πολιτική της συνοχής. Είναι ό,τι είχε πιο πολύ δυναμισμό στην υπόθεση στρατηγική Λισαβόνας. Τσέλερ, ε, συμφωνώ με, με την, την προσπάθεια της επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Τσέλα, να δούμε πώς θα έχουμε καινούργια άποψη αυτή τη στατική με την πολιτική της συνοχής και έτσι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το οποίο μας απασχολεί και εμάς και τις περιφέρειες. Αυτό το οποίο θέλουμε να το πετύχουμε και έτσι να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η ε, βεβαίω χρειάζεται κύριε Μποστινάρου, να έχουμε μια τέτοια πολιτική. Όντως θα πρέπει εδώ να δεσμευτούμε για πράγματα που δεν μας απασχολούν στην πολιτική της Λισαβόνας. Έχω να σας πω ότι όλα όσα είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όλα τα λαμβάνω υπόψη. Χέρι-χέρι θα βελτιώσουμε αυτήν την έκθεση και έχουμε μπροστά μα αυτή την περίοδο τη προθεσμίας των τροπολογίων, τόσο ώστε να κάνουμε ό,τι πρέπει. Η πρόεδρο. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, η προθεσμία όμω δεν είναι τόσο μεγάλη όσον αφορά τι τροπολογίε λόγω του Πάσχα. 24 Μαρτίου, 6 ώρα. Επομένω, προχωρήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε στι τροπολογίε σα. Έχουμε ακόμα κάτι που πρέπει να συζητήσουμε για ένα θέμα ουσίας. Η έκθεση Λάμπερτ Φανίστρ Ρόε. Πρόκειται για την έκθεση που αφορά την υλοποίηση των συνεργειών για κάποιες πολύ σημαντικές πολιτικές. Λάμπερτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. έχουμε ξεκινήσει από θέματα υψηλή πολιτική και πάμε τώρα σε κάποια πάρα πολύ πρακτικά θέματα, όχι τόσο υψηλή πολιτική. Είναι όμω πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, γιατί προσπαθούμε να δούμε οι πολιτικέ που ήδη τρέχουν πώ λειτουργούν στην πράξη. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη υπόθεση για την περιφερειακή πολιτική. Εδώ μιλούμε για συνέργειες, για περιφερειακό ταμείο, για ταμείο συνοχής, για έρευνα και ανάπτυξη για την κοινή αγροτική πολιτική, για την καινοτομία στις ΜΜΕ επίσης. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το χρήσιμο. Να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούμε επικοδομητικά από την Συναρμόδια Επιτροπή, την Ήτρε. Βέβαια, η συνεργασία ήταν πάρα πολύ αγαστή με την ε, Επιτροπή αυτή. Βγήκαν πολλές ιδέες στο προβληματισμό Και από εκείνους επίσης προέρχονται πάρα πολύ αξιόλογε ιδέες. όσον αφορά την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, στάθηκε δίπλα μου ως συνεισηγητής και αυτός επίσης συνέβαλε και τα είπαμε δύο φορές δύο ή τρεις φορές, λέει ο μιλητής, και νομίζω ότι καλά τα πήγαμε, γιατί μπορέσαμε να εστιαστούμε καλύτερα ε, στις ε, διάφορες επιμέρους δράσεις και δραστηριότητες. Τι έχουμε. Έχουμε πρώτα-πρώτα τους πόρους του 7ου προγράμματος πλαισίου και την ΚΑΠ. Και μπορείτε να δείτε πόσο έχει συμβάλει το Κοινοβούλιο στην διαμόρφωση αυτών. Έχουμε επίσης τον ξεχωριστό ρόλο του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με άλλη μεριά έχουμε τον ρόλο των κρατών μελών και τα κρατημέλη βέβαια θα βάλουν στις τελευταίες πινελιές δρώντας με τρόπο αποκεντρωμένο, με, την, με βάση την αποκέντρωση. Να δούμε πώς επομένως θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια πρακτικά μέσα πολιτικής. Και έτσι, αυτοί που είναι οι αποδέκτες αυτών όλων των προτάσεων, των ιδιών, των προγραμμάτων, που δουλεύουν επί τόπου, να μπορέσουν να ωφεληθούν. Να έχουμε κάποιες αρχές, κάποια εργαλεία που να μην χρειάζονται κάποιον ειδικό, κάποιον εμπειρογνώμονα να μην είναι περίπλοκα. Να είναι εύληπτα και σε περιφέρειες και σε πόλεις, γιατί αυτοί θα είναι οι αποδέκτες όλων αυτών. Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα πολιτικής που έχουμε. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να βοηθήσει και να επισημανθεί το τι πήγε καλά γιατί λιγότερο καλά. Περάσαμε από διαφορές φάσεις. Πρώτο πρώτα ήταν το non-paper της Κομισιόν, το έγγραφο του προβληματισμού. Μετέχαμε την ε, πράσινη βίβλο Μετά είχαμε τη διαπίστωση ότι πρέπει να ε, αναθεωρηθεί η κοινωνική πολιτική. Μετά είχαμε τον προβληματισμό για τα διορθωτικά ταμεία. Τώρα, με αυτή την έκθεση θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε και να δούμε ότι όλα έχουν την ε, εδαφική τους, την περιφερειακή τους πτυχή και να δούμε πώς να δουλέψουμε σε επίπεδο περιφέρειας. Να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε κάποιες ενέργειες ουσιαστικές και να έχουμε καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση αυτών των στόχων μεταξύ τους και βέβαια ανάπτυξη και έρευνα να πάει και αυτή στις περιφέρειες γιατί αυτό σημαίνει καινοτομία στα προϊόντα. Αυτό σημαίνει απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων. Έχουμε βέβαια κάποιες πόλεις, έχουμε κάποιους ε, θύλακες ούτως υπήν περιφερειών όπου μπορούμε να εστιαστούμε σε πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, οπότε να έχουμε ως πλεονέκτημα κάποιους τομείς αριστείας που ευδοκιμούν εκεί. Άρα, με σωστή αφετηρία, ας πούμε αν έχουμε για ενεργική πολιτική κάτι καλό, άρα σε μερικές περιφέρειες μπορούμε να δράσουμε ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα σημείο. Και αυτό θα γίνει με το, αν υπάρχει, με το να υπάρχει κάποια συνεργασία. Και έτσι και να συνεχίσουμε και παραπέρα. Άρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασία με την ε, Ήτρε. Και να κάνουμε την αξιολόγηση των ισχυουσών πολιτικών. Τώρα έχει ξεκαταστεί περισσότερο για το τοπίο της στατικής για το 2020. Όλα όσα μου είπαν οι συνάδελφοι ήταν ε, επίσης πολύ θετικό, επικοδομητική και η στάση των συνεργατών μας στην συνεργασία με την Ήτρε. και για την ΚΑΠ και για την έρευνα. Έχει σημασία το τι κάνουμε και άρα θα πρέπει να προσέξουμε όμως και, και την λίστα της ψηφοφορίας. Με μεγάλη μου χαρά τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη που είναι εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και μου, μου επιτρέπετε να μιλήσω σαν εισηγητή στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλνίστερ για την εξαιρετική πρωτοβουλία, διότι ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων στην Ευρώπη σπαταλάται, διότι δεν έχουμε την ε, σωστή κατεύθυνση για να προχωρήσουμε, άρα αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική. Πριν λίγο καιρό λάβαμε την Ατζέντα 2020 και τη συζητάμε. Ξέρουμε βέβαια ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν επέτυχε γιατί περιείχε πάρα πολλούς στόχους που δεν ήταν συγκεκριμένοι. Ενώ στη 2020 μπορούμε να επιτύχουμε 5-6 συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να μετρηθούν και μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία τους. Και χρησιμοποιώ χρησιμοποιώ την ε, νέα γερμανική λέξη streamlining, να τα κατευθύνουμε όλα προς μία κατεύθυνση ε, και ε, ίσως βέβαια δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη οι Υπουργοί Οικονομικών, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουν με ένα ποσοστό από το εθνικό ΑΕΠ και αν αυτό το επιτύχουμε δεν θα πρέπει να γίνει αυτό κατά τρόπον ώστε να συμβαδίζουν διαφορετικά εργαλεία τα οποία ενδέχεται να αντικρούονται και να ε, μην συμφωνούν. Πρέπει να ψάξουμε να επιτύχουμε ε, συνέργειες εδώ για την ηλεκτρική κινητικότητα παραδείγματος χάρη να ξέρουμε γιατί μιλάμε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ε, συζητήσει για τη τις ε, μπαταρίες ε, νικελίου ενώ εδώ και δύο χρόνια υπάρχει μία νέα κατεύθυνση ε, μπαταρίες λιθίου και η εξέλιξη προχωρά τρέχοντας. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην Ήπεθρο παραδείγματο χάρη όπου δεν υπάρχει υποδομή για να φορτίσουμε την μπαταρία ή αν δεν έχουμε ευρωπαϊκά πρωτόκολλα που να εξηγούν πώς μπορεί κανείς να μεταβεί από τη μία χώρα στην άλλη ε, τεχνολογικά. Και η Γενική Διεύθυνση έχει επιτύχει πολύ καλύτερη συνεργασία από ό,τι οι πολιτικές ομάδες και αυτό και με τον Λάμπερτ μπορέσαμε ε, να προχωρήσουμε από την ιδέα μίας ανακαλύψεως να δημιουργήσουμε ε, μία ροή η οποία προχωράει μέχρι την εφαρμογή με 5-6 φάσεις, με ενιαίες ε, δυνατότητες εφαρμογές, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο θα μπορούσε ήδη να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό. Αλλά χρειάζεται το πρόγραμμα SIP, η έρευνα, το Interreg, ε, δηλαδή περιφερειακό πρόγραμμα, ε, διάφορα σημεία. Διαφορετικά δεν θα πετύχουμε. Θα ήθελα στο μέλλον μία περιφέρεια να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα προγράμματα, αλλά υπάρχουν τρία προβλήματα. Αναφέρθηκα καταρχήν εις ε, τις διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής Δεύτερον υπάρχει ένα θέμα συγχρηματοδοτήσεως. Δεν μπορούμε ε, συγχρόνως ε, να ε, χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα από το Περιφερειακό Ταμείο και από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει όμως γιατί αν θέλουμε να βοηθήσουμε ορισμένες περιοχές Ευρώπης να ευθυγραμμιστούν χρειαζόμαστε άλλες μεθόδους. Και τέλος χρειαζόμαστε ειδικού οι οποίοι γνωρίζουν ε, αυτά τα τερπιτήπια, Δηλαδή χρειαζόμαστε καινοτόμο management. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, οι διαχειριστές να ε, επιμορφωθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ε, η, ηλεκτρική κινητικότητα που είναι πρωτοβουλία παραδείγματος χάρη της Ισπανικής Προεδρίας θεωρώ ότι είναι πολύ καλή πρόταση αλλά αν δεν το κάνουν οι Ισπανοί, έχει προτείνει ο κύριος Σταυρακάκης να γίνει στην χώρα τους. Δηλαδή ε, ε, υπάρχουν δυνατότητες ανακατανομής ε, των διαφόρων ταμείων, συνοχής, περιφερειακό κτλ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν επικοδομητικά. Να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές καινοτομία, έρευνες που επιτρέπουν να προοδεύσουμε διαφορετικά. Θα βρισκόμαστε είμαστε μονίμως σε μία άτακτη κατάσταση. Έχουμε την κατάσταση της Ελλάδος αυτή τη στιγμή σαν ένα παράδειγμα. Σε λίγο έρχεται η Ισπανία, η Πορτογαλία, θα υπάρξουν πολλοί. Άρα χρειάζεται ε, μία πρωτοβουλία σαν του κυρίου Βανίστελ Ρόι που συμβάλλει πολύ επιτυχώς στην ατζέντα του 2020 διότι διαφορετικά δεν θα αντεπεξέλχομαι. Ευχαριστώ. Ε, ο Μίχαλ Χόγερ τώρα που είναι σκιώδης συγητής. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές ε, μας ε, μίλησαν ε, για αυτά τα θέματα, τα συζητήσαμε ήδη. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Γιάνν Βαλίστερ Ρόι για την πρωτοβουλία του και τον Γιώργο Χατζημακάκη, τον συνάδελφο από την Επιτροπή Ήτρε και θα περιοριστώ σε λίγα σχόλια τώρα. Διεφάνει σαφώς πού υπάρχουν συνέργειες για το μέλλον, πού μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα μεταξύ ε, ερευνητικών προγραμμάτων και μεταξύ ταμείων ε, συνοχής ε, και διαρθρωτικού και ε, συγχρόνως υπάρχει μια καλή βάση για να υπάρξουν διάφορες εφαρμογές αφενός top down από πάνω προς τα κάτω ευρωπαϊκή πολιτική ε, διεθνής πολιτική βασική έρευνα και δίκτυα και υπάρχει συγχρόνως ανάγκη να μπορέσουμε να βρούμε μια θέση για το αντίθετο δηλαδή την προσφορά από κάτω προς τα πάνω διότι για διάφορα πράγματα υπάρχουν απαιτήσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για μικρομεσαίες σχολές οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται διότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια, διότι η έρευνά τους δεν είναι τόσο επαναστατική όσο θα χρειαζόταν και ε, όπου ε, στα πλαίσια του Ίντερεκ χρειάζεται τεράστια συνεργασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά ε, στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας όσον αφορά τα clusters στον περιφερειακό τομέα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι προς όφελος και των περιφερειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή και αυτό είναι το κέρδος μας επί του προκειμένου ότι ο κύριος Βανίστελ Ρόι και ο κύριος Χατζημαρκάκης έχουν εκπονήσει ένα ε, σύνολο το οποίο παρουσιάζει τα σημεία τομής ε, και είναι πολύ σημαντικό διότι έτσι ε, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα αναμείνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση ε, στα έγγραφα, στις διαδικασίες, όλα αυτά να απλοποιηθούν, να διατυπωθούν ενιαία και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ακόμη περισσότερο είναι στο μέλλον να υπάρχουν δύο οδοί. Μία από πάνω προς τα κάτω για την προώθηση της έρευνας αλλά όπου και οι περιφέρειες κατά προτίμηση ενιαία θα μπορέσουν να προωθήσουν τις ε, περιφερειακές οι ιδιομορφίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Είναι θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε καθόλου εδώ. Δεν ξέρουμε που υπάρχουν δυνατότητες καινοτομία και θα πρέπει να αφήσουμε και στους μικρούς τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να απαιτήσουμε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Ε, νομίζω ότι είμαστε γενικά στο σωστό δρόμο δρόμο. Θα χρειαστούν ε, μικροπροσαρμογές όπως είπα γενικώ, αλλά η γενική γραμμή νομίζω ότι είναι ικανοποιητική σε αυτό το σημείο ε, και τουλάχιστον ε, η πρωτοβουλία της ομάδος των φιλελευθέρων πρέπει να τύχει συγχαρητηρίων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Φανιστερό για την εκθεσή του αλλά και τον συνεισηγητή για όλε τι ιδέε του. Εγώ τώρα έχω τι εξή παρατηρήσει που θα τι κάνω και ω τροπολογίε. Πρώτα-πρώτα νομίζω ότι θα πρέπει η έκθεση αυτή να προσέξει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα είναι η προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Σημαντική αύξηση των πόρων για την καινοτομία όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εξοικονομική ενεργείας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και επίσης να έχουμε καλύτερες συνεργειακές επιδόσεις των κτηρίων τόσο ώστε να ε, προγιάνουμε το έδαφος για την ε, σχετική οδηγία η οποία οδηγία σύντομα πρόκειται να εγκριθεί στο Κοινοβούλιο. Επίσης πρέπει να τονίσω στην εκθέση αυτή το ότι δεν έχει επισημανθεί η σχέση μεταξύ καινοτομία και κοινωνικής ένταξης γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την συνοχή με την ανταγωνιστικότητα μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής πολιτικής ακριβώς όπως και στο κοινωνικό πρόγραμμα in Europe. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει την ε, ανάπτυξη, στην ε, καινοτομία σε κάποιες περιοχές μη προνομιούχες τη ευρωπαϊκή πόλη και κατά αυτόν τον τρόπο συγκεράζονται περισσότεροι στόχοι. Δηλαδή πρώτα-πρώτα έχουμε ε, κάποια ε, κατάρτιση σε αυτές τις ε, φτωχές γειτονιές, ε, να γεφυρωθεί το χάσμα ε, στις κοινωνικές ανισότητες σε πόλεις και περιφέρειες, να βελτιώσουμε την κινητικότητα σε σχέση με τις πόλεις και τις υποδομές, επίσης να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων των πόλεων, η ατμόσφαιρα, ε, η καταπολέμηση του θορύβου συγκεκριμένα επίσης, το πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση στην απασχόληση οι νέοι. Κάτι το οποίο περνάει μέσα από την αναβάθμιση της κατάρτισης και της ευκολίας πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Επίσης, τονίζει η έκθεση το ότι χρειάζεται να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών κοινοτικών προγραμμάτων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Θα πρέπει αυτή η έκθεση να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσει την κατάρτιση στους ε, τοπικούς, στις τοπικές, και έτσι να μπορούμε να έχουμε ε, μια μεγαλύτερη ε, πρικοδότηση και συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε έξι ομιλητέ. Παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Εγώ θα ήθελα αν μπορώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βανίστερ Ρόι διότι μίλησε για την συνέργεια στην έρευνα και ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Περίοδα 2007-2013, μεταξύ του 2000 και του 2013, ε, έχουμε τριπλασιάσει ε, την ε, χρηματοδότηση για την καινοτομία και την ανάπτυξη και την έρευνα αλλά αυτό μόνο σε σύγκριση με την προηγούμενο περιοχή, δηλαδή 50 εκατομμύρια ε, χρησιμοποιήθηκαν για την ε, καινοτομία και την έρευνα. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα προς τα εμπρό σε σχέση με το παρελθόν, αλλά αν συγκρίνουμε με την Κίνα και ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να πούμε ότι είναι απλώς ένα πρώτο βήμα και πρέπει να προχωρήσουμε διότι βλέπουμε πώς θα πρέπει να πάμε προς τα εμπρός. Ε, έχω να κάνω ελάχιστες παρατηρήσεις. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τα πρότυπα επιτυχία στα πλαίσια του τριγώνου που αποτελούν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές. Καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να προέρχονται από, τις, ε, ε, ε, από τα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να προωθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές. Και διαπιστώνω με τα χαράς ότι εδώ θεωρούμε ότι ε, η πολιτική θα συμβάλλει πάντοτε στην επίλυση των βασικών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, των διαφορών μεταξύ ε, των διαφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού των δημογραφικών ε, και κλιματολογικών αλλαγών εξετίμησα ιδιαιτέρως τη δυνατότητα που υπάρχει να προτείνουμε διάφορα εναύσματα για να εφαρμοστούν μέτρα καινοτόμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει πιο σημαντική στήριξη ε, για τις πολιτικές οι οποίες προωθούν τις συνέργειες ε, για την ε, καινοτομία και την δημιουργία θέσεων εργασίας όπως άλλωστε το αναφέρει ο εισηγητής το τέλος εκθέσεως και τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Βανίστελ Ρόι για αυτή την έκθεση διότι ανοίγει νέους δρόμους και κάνει μία πολύ συγκεκριμένη ανάλυση διαφόρων πολιτικών και πιστεύω ότι αυτή η οδός θα πρέπει να προωθηθεί και να συνεχίσει να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, οι οποίες θα μας δείξουν πόσο ε, μπορούμε να επιτύχουμε και άλλωστε συνάδελφοι πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι στην Επιτροπή μας για Περιφερειακή Ανάπτυξη είμαστε μια εγκάρσια έκθεση και με τη συνθήκη της Λισαβόνας συμμετέχουμε ακόμη πιο ενεργά στη λήψη των αποφάσεων. Ε, χρειάζεται λοιπόν να συγκεράζουμε τις διάφορες απόψεις. Είναι κάτι το οποίο τονίζουμε συχνά διότι όλοι θα θέλανε να βάλουν χέρι στο καζάνι της πολιτικής συνοχής ε, αλλά νομίζω όπως άλλωστε το έπραξε και ο Λάμπερτ Βανίστελ ότι πολλοί σωστά πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο, άρα εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Και ε, γυρίζω τώρα προς ε, τον ε, εισηγητή της Επιτροπής Ήτρε, τον κύριο Χατζημαρκάκη, που λέει ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε, Αν θέλουμε η καινοτομία να στηριχθεί και ε, οικονομικά και να χρησιμοποιηθεί ε, και στις περιφέρειες που μπορούν να αναλάβουν δράση. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω να παραπέμψω σε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2009 που αναφέρεται ε, για την μετάβαση προς μία εποχή της, της αλλαγής όπου μιλά για την προώθηση των καινοτομιών ή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι στο έγγραφο αυτό βασίζεται η έκθεση του συναδέλφου Βίνκλερ για να υπάρχει η επαφή. Δηλαδή ότι θα έχουμε επιτύχει από τις εκθέσεις Βανίστελ Ρόι και να συντονιστούν για να μπορέσουν να διατυπωθούν και να περιληφθούν στην έκθεση για την καινοτομία και την έρευνα. Ευχαριστώ. Η Σόφη και μετά ο κύριος Αγκουράκης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση του Λάμπερτ Βαντιστερό είναι εξαιρετική και δεν νομίζω πως έχουμε πολλά πράγματα, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Όλα λαμβάνονται υπόψη, επικοινωνία, καλές πρακτικές, ε, τα βασικά προγράμματα είναι καλά στοχευμένα κτλ. Το μόνο σημείο που εγώ θα ήθελα να θίξω είναι η σημασία της πολιτικής συνοχής και των διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί η Ευρώπη στις περιοχές μας. Συμφωνούμε και διαπίστωσα στη Γαλλία εγώ μάλλον υλοποίησα στη Γαλλία μια ανέκθεση για τους λόγους για τους οποίους αυτές οι πολιτικές και αυτά τα προγράμματα δεν ε, τα έχουν ιδιοποιηθεί οι τοπικοί φορείς και γιατί τελικά αυτές οι πολιτικές και αυτά τα προγράμματα διατηρούν ε, μια εικόνα δεσμευτική και δύσκολη, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω πως ε, ο λόγος για τον οποίο οι διάφορες αυτές πολιτικές δεν εφαρμόζονται με το δυναμισμό και τη δυναμική που θα θέλαμε να δούμε στα, στις περιοχές μας προκύπτει από την περιπλοκότητα της διαδικασίας. Αυτή η πρωτοβουλία της ε, συνεργίας, συνέργειας μεταξύ πολιτικών και προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική, κυρίως σε κρίση όπως αυτή που διανύουμε σήμερα. Και είναι πάντα δύσκολο γιατί αυτά προτίθενται γιατί προστίθεται το ένα στο άλλο, η διαχείριση δηλαδή των προγραμμάτων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία και στην εφαρμογή, συντονισμός στην εφαρμογή των διαφόρων αυτών πολιτικών μέσω μιας απλοποίησης των διαφόρων διαβημάτων, κυρίως για τα έγγραφα, έχετε δίκιο, που θα πρέπει οι διάφοροι φορείς να συμπληρώνουν, ε, για να, που θα πρέπει να είναι τα ίδια για όλα αυτά τα διαβήματα. Πρέπει να απλοποιήσουμε, γιατί από αυτό εξαρτάται η εικόνα της ε, πολιτικής συνοχής και των διαφόρων προγραμμάτων και εξαρτάται και η εικόνα της Ευρώπης από αυτό. Πιστεύω πως θα πρέπει δηλαδή να επικοινωνήσουμε, να προχωρήσουμε προς μια διαφάνεια, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε μέσα σε ένα, πνεύμα απλοποίησης, ώστε όλα αυτά να είναι αποτελεσματικά και να δώσουμε μια μια θετική και δυναμική εικόνα σε όλες αυτές τις πολιτικές και τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαγκουράκης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι το εξή. Θα πω κάποια πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την προσπάθεια του εισηγητή, η οποία είναι σοβαρή και σωστή. Ε, εγώ καταλαβαίνω και από το κείμενό του υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του επιστήμονα και του πολιτικού. Και θα σας πω τι εννοώ, επιτρέψτε μου λιγάκι να πάμε λίγο στην βασική έρευνα. Ε, ο κύριος ε, εισηγητής κάνει λόγο για το ότι στα περιφερειακά προγράμματα δαπανήθηκαν 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι μας, μπορεί να δαπανήθηκαν τόσα και πολύ περισσότερο, αλλά κανείς, ούτε στις ΗΠΑ, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Κίνα, δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την τεράστια οικονομική κρίση που ξέσπασε πριν δύο χρόνια. Η οποία οικονομική κρίση βεβαίως έχει κοστίσει ε, τόσα πολλά πράγματα σε πολλές χώρες, σε πολλούς λαούς και κυρίως στους εργαζόμενους. Το λέω αυτό κυρία Πρόεδρε διότι ε, όσα δισεκατομμύρια για να ξοδέψουμε ε, δεν θα σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων και στο ύψος των αναγκών των σημερινών διότι όλα αυτά εξυπηρετούν δυστυχώς μια κοινωνία που έχει ως στόχο την ανταγωνιστικότητα και το κέρδος. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε με την στρατηγική της Λισαβόνας το ίδιο και χειρότερο θα γίνει στο μέλλον αν δεν αλλάξουν οι προτεραιότητε. Και σα έφερα αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όταν ξοδεύονται δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων σε τόσε χώρε ώστε το πιο σημαντικό, το πιο βασικό ζήτημα που μα απασχολεί όλου, να μην μπορέσει να το έχει προβλέψει κανεί. Έτσι θα πάμε. Δεύτερο ζήτημα, το κάνω λίγο πιο ειδικό όσον αφορά την Επιτροπή μα. Αν έχω καταλάβει καλά, ο ρόλο τη επιτροπή μα είναι να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των περιφερειών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή οι περιφέρειες όσο γίνεται περισσότερο να συγκλίνουν. Αν δούμε όμως ε, και την προηγούμενη έκθεση και το σημείο 13 της έκθεσης ε, που συζητάμε σήμερα, τα πράγματα μπαίνουν ακριβώς ανάποδα. Δεν είναι δηλαδή τι θα πάρουμε από τη στρατηγική του, του 2020 για να προωθήσουμε τη συνοχή δεν ήταν τι θα πάρουμε από τη στρατηγική της Λισαβόνας για να προωθήσουμε τη συνοχή, αλλά πάει ανάποδα. Πώς η πολιτική της συνοχής θα εξυπηρετήσει τη στρατηγική του 2020. Αν πάμε έτσι Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, το βέβαιο είναι ότι οι διαφορές θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλες. Και θα γίνουν πιο μεγάλες οι διαφορές γιατί. Γιατί η στρατηγική του 2020 είναι ακριβώς η ίδια με αυτή της Λισαβόνας. Ανταγωνιστικότητα. Από αυτή την άποψη όλα τα ερευνητικά προγράμματα θα εξυπηρετούν τον στόχο της ανταγωνιστικότητας και θα πηγαίνουν βεβαίως σε εκείνες τις περιοχές και σε εκείνα τα πανεπιστήμια που είναι πιο ανταγωνιστικά. Γιατί να πάνε ας πούμε στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές από τη στιγμή που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα το στόχο της ανταγωνιστικότητας. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα, υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν μηχανισμοί που να ανεβάσουν το επίπεδο της περιφέρειας. Και τελειώνει, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στόχος μας η δημιουργία πολλών Silicon Valley στην Ευρώπη. Εξάλλου αυτό το μοντέλο έγινε και πριν τα 20 ε, χρόνια, που περάσαμε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ε, ξέρουμε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα κριτήρια και κάτι προσπαθεί να πει ο κύριος ε, ε, εισηγητής στην, ε, έκθεσή όταν λέει θεματική εστίαση ενάντια εδαφικής στο σημείο σίγμα ταφ της έκθεσης. Πραγματικά, ποια είναι αυτή η θεματική εστίαση. Για τα ζητήματα αυτά όμω δεν υπάρχουν ε, πώς το λένε, στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο λέω η έκθεση κάνει μια προσπάθεια όμω δεν αντιμετωπίζει το κύριο ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Very much. And before I ask again... Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν να δώσω και πάλι το λόγο στον ε, Βανίστερόι, θα δώσω στον Μικέλ Ανταμπάς από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Region. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα πρέπει να πω ότι πρόκειται για ψηλής ποιότητα στροφή για σκέψη. Είναι πολύ ευπρόσδεκτη η εκθέση αυτή και μας δίνει δύο βασικά θέματα, τουλάχιστον δύο για να τα σκεφτούμε. Το ένα είναι σαφώς το πώς θα συγγραμμιστεί η πολιτική συνοχή με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 μέσω των όσων αποκαλούνται στην έκθεση ε, ενισχυμένη earmarking και θεματική η στόχευση. Το δεύτερο είναι η σαφής αναγνώριση πως η αριστεία στην έρευνα και η περιφερειακή καινοτομία είναι συμπληρωματικά και χρειάζονται. Και η σύνδεση ανάμεσα στα δύο είναι πιθανόν αυτό που εκείνο αποκαλεί ευφύ, πράσινη, περιφερειακή ειδίκευση. Αυτό σημαίνει πως η ευρωπαϊκή Κομισιόν θα πρέπει να φτιάξει κάποιε επιλεγμένες προτεραιότητες για τις καινοτομίε και περιφέρειες ανάλογα με τι δυνατότητε του να ευθυγραμμιστούν μέσω των πολιτικών με αυτές τις πιο το πιο γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα ήθελα τώρα να κάνω δύο συγκεκριμένα σχόλια για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με, αυτές τις, με αυτό το συντονισμό ε, καταρχήν όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ των συστημάτων στην Κομισιόν για αυτά τα δύο είδη Ε, κενή διαχείριση, προγράμματα και επικουρικότητα. Το άλλο είναι η άμεση διαχείριση που βασίζεται σε ανταγωνισμό και προγράμματα, συνήθως προγράμματα διεθνούς φύσης. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, είναι δύο διαφορετικές ε, διοικητικές κουλτούρες για τους διαφορετικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσει κανείς τα χρήματα. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν από τα μέσα του δεκαετίας του 90, από την πρώτη φορά που φτιάξαμε ένα χάρτη συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσει, ξεκινήσαμε την ε, περιφερειακή στρατηγική συνεργασία. Έχει, δια... έχει διαρκέσει 10 χρόνια και θεωρήθηκε από διάφορους φορείς ως επιτυχής. Πέρυσι για δεύτερη φορά υπογράψαμε ένα χάρτη συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις ΓΔ και εργαζόμαστε για δύο συγκεκριμένα προγράμματα από το, πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο. Το ένα είναι η Μεγάλε μεγάλες υποδομές και ανάπτυξη και το άλλο είναι το δυναμικό, το ερευνητικό και προσπαθούμε να αλληλοϊποστηριζόμαστε. Το άλλο που, σας, που αναφέρθηκε ήταν η διάδοση των καλών πρακτικών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μέσω τη πρωτοβουλία για τι ε, περιφέρειες και την οικονομική αλλαγή Έχουμε προγράμματα από 10 με 15 περιφέρειες, τις οποίες χρηματοδοτεί η ΓΑΜΑ και να σας θυμίσω τέλος ε, τι σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές, την απλοποίηση που εφαρμόστηκε πέρσι στους κανονισμούς μας σε σχέση με τα σε, ε, <coughs> καταποκοπή ποσά για το υπερκόστος και επίσης ε, το κόστος κλίμακας και τις προσπάθειες που έγιναν πέρυσι για ευθυγράμμιση. Ευχαριστώ. Ο κ. Φανέστελ Ρόι δεν είναι υποχρεωτικό, αν δεν θέλετε, ναι, είναι ευχαρίστω να κάνω δύο τελικέ παρατηρήσει Κάποια από τα σχόλια που έγιναν. είναι πως ε, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να αναζητήσουν την αριστεία στα ερευνητικά προγράμματα. Δεν είναι λάθος κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Πρόκειται για μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και ένα απαραίτητο θέλουμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Θα πρέπει να έχουμε διάφορα ταμεία γιατί μέσω της περιφερειακής πολιτικής μπορούμε στην πράξη να εφαρμόσουμε αυτό που κάνει το Ταμείο Έρευνας και Καινοτομίας όσον αφορά την οικολογία, όσον αφορά την ενέργεια, και όσο αφορά την ε, κοινωνική καινοτομία. Και πώς μπορούμε τώρα όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Ε, την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, μάλιστα τώρα, τότε την εβδομάδα, υπήρξε μια, ένα συνέδριο με 500 συμμετέχοντες. Ήταν η εβδομάδα των καινοτόμων περιφερειών και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν παρόν, υπήρξε μέγας ενθουσιασμός και φαίνεται ότι στην πράξη ασχολούμαστε με τον εντοπισμό της αριστείας για προγράμματα που συνδυάζονται με την ερευνητική υποδομή. Αυτά όλα λοιπόν είναι δυνατόν να γίνουν, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για να χρηματοδοτηθούν οι ερευνητικέ δομές. Οι εμπειρογνώμονες του τομέα το λένε ότι πρόκειται για πράγματα βεβαίως που δεν γίνονται εύκολα, αλλά πρέπει να γίνουν με αυτόν τον τρόπο γιατί υπάρχει μια λογική οι πολιτικοί ηθήνοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν στα επόμενα χρόνια και αν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα 20 χρόνια θα πρέπει να γνωρίζουν τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουν και να τις κάνουν. Ήδη υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι έτοιμες να επενδύσουν όπως και τα κράτη-μέλη το ίδιο. Ακριβώς όσον αφορά την ε, το περιφερειακό επίπεδο, νομίζω πως η έκθεσή μου συμβάλλει στο να γίνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το τομέα. Η θεματική επιλογή υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ε, συγγνώμη, προτεραιότητες και αυτές μεταφράζονται σε ε, πρωτοβουλίες της ίδιας της περιφέρειες. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχει μόνο μια ιονή αντίφαση, η οποία όμως δεν είναι αληθινή στην πραγματικότητα. Τα κονδύλια για την έρευνα έχουν διπλασιαστεί, αλλά εμείς πρέπει να ανταγωνιστούμε τη ΣΥΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, Άρα, τα περιφερειακά ταμεία μπορούν να μεταφραστούν σε καινοτομία στις περιφέρειες. Και με αυτόν τον τρόπο οι δυνατότητες μας αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι ένας από τους πυλώνες που οδηγούν στην ανταγωνιστικότητά μας. Περιφερειακοί ηγέτες και τέρι πρόεδροι των περιφερειών, ε, δήμαρχοι, Όλοι αυτοί προβαίνουν σε επιλογές, δεν κάνουν όλα τα ίδια πράγματα, οπότε πρέπει να υπάρχει μια θεματική επιλογή. γιατί στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο διαφοροποίησης στις περιφέρειες και η συγχρηματοδότηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Ναι, η κοινωνική διάσταση την έχουμε λάβει υπόψη. Μπορούμε ίσως να βελτιώσουμε τις ε, τροπολογίες. Η βιωσιμότητα βεβαίως ναι, επίσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς αυτό. Θα εργαστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα στο να σας δώσω και το κείμενο. 24 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, όπως είπαμε. Θα ήταν ωστόσο καλό να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση για τη στρατηγική 2020, έτσι ώστε δηλαδή τα μέσα αυτά να υποστηρίξουν τη διατήρηση αυτών των στόχων. Να αναφέρουμε άλλη μια φορά την ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν 24 ή όχι. The for Ναι, η προθεσμία αυτή είναι 6 ώρα της 24 Μαρτίου. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστούμε τους ε, συνεισηγητές. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία Χατζημαρκάκη και Φανή Τελρόη και η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τώρα. Το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε είναι η ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις των συντονιστών, τις χθεσινές τους αποφάσεις γιατί είχαμε αυτή την ε, απόφαση όσον αφορά το πού θα πάει η γνωμοδότηση για την ε, πολιτική για την θάλασσα Οργανώθηκε επίσης ε, αυτό το εργαστήρι για την απλούστευση της ε, νέας πολιτικής συνοχής το 2013. Οι δε συντονιστές συμφώνησαν ε, στις 25 Μαρτίου, μέχρι τις 25 Μαρτίου να έχουν στείλει παρατηρήσεις και ερωτήσεις, ό,τι θέλουν να συζητηθεί κατά το εργαστήρι. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνει αποστολή στη Ρουμανία για τρεις μόνο μέρες και μας υποσχέθηκαν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό στην από τη Ρουμανία, μείνει ε, ακρόαση όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση για την περιφερειακή μας πολιτική, κάτι που θα λάβει χώρα τους αμέσως επόμενους μήνες ή μήνα. Επίσης, γνωμοδότηση τον τρόπο τέλο πάντων που θα, θα κινηθούμε όσον αφορά την πολιτική της καινοτομία. Που για άλλη μια φορά θα είναι συνεργασία με την κυρίω αρμόδια Ήτρε. Πιέζει όμω ο χρόνο, οπότε δεν θα γίνει γνωμοδότηση. Όμω θα συντάξουμε μια επιστολή την οποία θα προετοιμάσει η γραμματεία και στη συμφωνήθηκε ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Αυτά αποφασίστηκαν χθε από τους συντονιστέ. Το τελευταίο τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι τόπος και χρόνος της συνειδήσης που το ξέρετε, Δευτέρα 26 του μηνός και Τρίτη 27 Απριλίου. 3 με 6,5 τη Δευτέρα, 9 με 12,5 την Τρίτη. Είχαμε πάρα πολλά θέματα, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε πολύ σημαντικέ εκθέσει. Όμω, τα συζητήσαμε όλα πολύ καλά Ευχαριστώ που ήσασταν όλοι προετοιμασμένοι. Ευχαριστούμε όλους, αλλά και τους διερμηνείς μας. Για τα όσα κάνουμε αυτές τις ε, δύο μέρες. Πέρα συνδυάσεως.